Θέλετε να αρχίσουμε σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να καθίστε. Συνήθως ε, Ε, αναμεταδίδεται μέσω ίντερνετ ε, η συνεδρίασή μας οπότε σας παρακαλώ να προσέχετε όταν μιλάτε. Λοιπόν, η ημερήσια διάταξη, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Ελπίζουμε να αντιστρέψουμε τα δύο σημεία σχετικά με την ακρόαση και την έκθεση ΚΡΕΛ αλλά δεν μπορώ ακόμη να σας εξαγγείλω τίποτα. Να είστε έτοιμοι. Τώρα, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια στην ημερήσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 2 που είναι οι ανακοινώσει τη Προέδρου. Έχω μόνο 2-3 σημεία αρκετά σύντομα να σας αναφέρω. Έγινε όπως ξέρετε η συνεδρίαση των Υπουργών για την Πολιτική Συνοχή στις 22 Νοεμβρίου στην Λιέγη. Συμμετείχα ως πρόεδρος, καθώς επίσης και ο κύριος Βανίστελ Ρόι, στη Λιέγη πάλι. Τα βασικά θέματα ήταν το μέλλον της πολιτικής συνοχής με ιδιαίτερη διασύνδεση με την Ευρώπη του 2020 η μεταρρύθμιση της πολιτικής όπως ε, περιλαμβάνεται στην πέμπτη έκθεση συνοχής και καθώς επίσης και για τα διάφορα θέματα αιρεσιμότητας. Και οι δύο ομιλίες σας έχουν διανεμηθεί και αμέσως μετά από την συνάντηση αυτή σας είχαμε διαβιβάσει τα απορίσματά της τα οποία νομίζω είναι τέτοια που αποδίδουν καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για το προσεχές μέλλον και που κατά τη γνώμη μου ε, αξίζει να αναγνωστούν από όλες και όλους. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη ανακοίνωση, αναφέρεται στην συνάντηση συντονιστών του Στρασβούργου στις 24 Νοεμβρίου σημαντική συνάντηση διότι αποφασίσαμε σε αυτήν να κατανείμουμε πρόσθετους βαθμούς στις πολιτικές ομάδες. Οι συντονιστές λοιπόν απεφάσισαν να δώσουν σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ρέτζι δύο πρόσθετους βαθμούς. Η συμφωνία υποστηρίχθηκε από το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές, τους Φιλελευθέρους ενώ αντίθετη ήταν της Ενωτικής Αριστεράς και των Πράσινων η οποία ομάδα των Πράσινων εξέφρασε επιφυλάξεις επί της αποφάσεως και δήλωσε ότι θεωρεί ότι έτσι αλλάζουν οι κανόνες του συστήματος TONT. Βέβαια η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν συμβαίνει αυτό. Το εξετάζουμε πάντως. Επίσης στις 30 Νοεμβρίου είχαμε συνάντηση όπου πάλι τέθηκε θέμα από τον κύριο Βανίστελ Ρόι για, σχετικά με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 50 για εκθέσεις για την νομοδοτήσεις μάλλον για την Επιτροπή Θεμελιτών Ελευθεριών για τους Ρώμα κλπ. Αυτά θα τα δείτε και τα πρακτικά της συναντήσεώς μας. Επίσης, συζητήσαμε την κατανομή εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων και ιδίως για θέματα μεταρρυθμίσεως της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, την ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την έκθεση την ανέλαβε, την γνωμόδοτηση την ανέλαβε το Λαϊκό Κόμμα και για την νομοθεσία μετά από το 2013. Σήμερα θα παρακαλέσουμε να λάβει το λόγο ο Επίτροπος Χάν για δύο θέματα που είχαμε θέσει στη συνάντησή μας. Αφενός την ανάγκη ξεχωριστής νομοθεσίας για το Περιφερειακό Ταμείο και για το Γεωργικό Ταμείο, καθώς επίσης θα ρωτήσουμε τον Επίτροπο σήμερα σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής του στρατηγικού πλαισίου από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διαταξή μας ήταν η συμφωνία συστάσεως των συντονιστών σχετικά με τις ε, συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια του χρόνου. Θέλουμε να διεξαχθούν οι συναντήσεις αυτές, η συνάντηση μάλλον αυτή, οπότε συμφωνήσαμε ότι θα γίνει από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τώρα οι συντονιστές να αποφασίσουν επί του θέματος και του χρονοδιαγράμματος. Θέλουμε επίσης τρεις μήνυα ακροάσεις του χρόνου μία για την ισότητα των φύλων στην πολιτική συνοχή, δεύτερο η πολιτική συνοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτο συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και γενικά πολιτική γειτονίας και πολιτική απέναντι στις υποψήφιες χώρες και βέβαια τον ρόλο της πολιτικής συνοχής σε, όλα, σε όλες τις σχετικές πτυχές του θέματος αυτού. Θα γίνουν λοιπόν αυτές οι μήνυα ακροάσεις ε, του χρόνου όταν θα έχουμε πλέον στα χέρια μας το χρονοδιάγραμμα. Συζητήσαμε και τις εξωτερικές μελέτες για το 2011 μέσα στα πλαίσια δηλαδή της ε, μακροοικονομικής συνοχής για να κατανοήσουμε τη νομική βάση αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτά συνοψίζουν τα όσα συζητήσαμε και αποφασίσαμε στη διάρκεια των συναντήσεων. Εδώ λήγουν οι ανακοινώσεις μου. Εάν δεν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση του Επιτρόπου Χάν τον οποίο ευχαριστώ για την έλευσή του. Κύριε Πίτροπε, θα θέλαμε να ακούσουμε, επειδή και εσείς ο ίδιος προτείνατε, ε, μάλλον εξέ, ε, εκδώσατε την έκθεση για την, την πέμπτη έκθεση συνοχής και τη στρατηγική του Δούναβη. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και τα δύο αυτά θέματα. Παρακαλώ τους συναδέλφους μου να είναι το δυνατόν σύντομοι <clears throat> μετά στις τοποθετήσεις τους και στις ερωτήσεις τους, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Επίτροπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Είχαμε την ευκαιρία αμέσως μετά την λήψη αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είχαμε λοιπόν ήδη την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση συνοχής και ιδίως τα απορίσματά της. Είναι σημαντικό να σας εξηγήσω και τι έγινε τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το θέμα αυτό. Όπως είπε ήδη η κυρία Χιούπνερ, σας μίλησε δηλαδή για τον επίσημο ή το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, όπου η σχετική έκθεση ήταν αντικείμενο της συζητήσεως. Στο μεταξύ είχα την δυνατότητα στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να μιλήσω για την απαλλαγή του 2009 το θέμα ετέθηκε σχετικά με το μέλλον και νομίζω ότι συνολικά προσβλέπουμε σε μια καλή εξέλιξη του δημοσιονομικού ελέγχου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Τανούτα Χύπνερ ως πρώην επίτροπο και βεβαίω ε, την υπηρεσία, αλλά και τις περιφέρειες οι οποίες έχουν καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες μέσα στα πλαίσια του shared management. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια πλέον και να επαναπαυθούμε στις μέχρι τώρα δάφνες μας. Ελπίζω το έτος 2009 να επαναληφθεί και το 2010. Είναι σημαντικό να τονίσω και εδώ μπροστά σας ότι το 2009 σε ό,τι αφορά το δείγμα το οποίο έλαβε το ελεγκτικό συνέδριο δεν ήταν απλώς τυχαίο και τυχερό, διότι θα είδατε ότι συνολικά εξετάστηκαν 15 χώρες. 180 έργα σε 15 χώρες. Και μεταξύ αυτών και χώρες που είναι γνωστές για το γεγονός ότι σημειώνονται εκεί προβλήματα και στον δημοσιονομικό έλεγχο και έχουμε κάνει και το λεγόμενο risk monitoring και αρχίζουν λοιπόν και φαίνονται τα αποτελέσματα. Και εν προκειμένου ίσως είναι σημαντικό να πω ενώπιον σας ότι ο μηχανισμός που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνεται στους νέους κανονισμούς δηλαδή η δυνατότητα διακοπής πληρωμών ήδη στην περίπτωσή μας μπορεί να επιβληθεί από το Γενικό Διευθυντή της DG Regio. Και ο μηχανισμός αυτός έχει αποδώσει. Ως πρώτο βήμα, ως πρώτο μέτρο είναι η διακοπή και μετά, εάν αυτό δεν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, υπάρχει η δυνατότητα, δηλαδή η διακοπή μπορεί να διαρκέσει maximum 6 μήνες, μετά είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε μία καταρχήν αορίστου χρόνου αναστολή. Πέρσι κάναμε 7 τέτοιες αναστολές. Σήμερα έχουμε 43, μέχρι σήμερα 43 διακοπές και νομίζω 16 από αυτές τις διακοπές ισχύουν ακόμη. Ο, ο μέσος χρόνος διάρκειας των διακοπών αυτών είναι των τριών μηνών και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία αναστολή suspension. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι ο μηχανισμός αυτός αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα. Νομίζω ότι μπορούμε αλλά και πρέπει κιόλας διότι την εντολή αυτή μας έχει δώσει το Κοινοβούλιο στην επόμενη προγραμματική περίοδο να εγγύψουμε περισσότερο στα αποτελέσματα, στην αποτελεσματικότητα δηλαδή της πολιτικής λαμβάνοντας ως βάση τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 που νομίζω ότι αυτή είναι ακριβώς που θα αποδείξει ότι χρειαζόμαστε μια περιφερειακή πολιτική που οφείλει να λάβει υπόψη τις ανάγκες όλων των περιφερειών ώστε να μειωθούν οι αντιθέσεις στο βιωτικό επίπεδο, στο επίπεδο ευημερία, στην οικονομική απόδοση και το καθεξής. Το δεύτερο μέτρο βέβαια είναι η ευρωπαϊκή πολιτική να προάγεται με έργα στις περιφέρειες και να καθίσταται σαφές ότι οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρώπης του 2020 μπορούν να υλοποιηθούν. Διότι πώς θα γίνει η καταπολέμηση της φτώχειας εάν δεν γίνει προσπάθεια ταυτόχρονα σε όλες τις περιφέρειες. Πώς θα αυξήσουμε αυτούς που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, πώς θα αυξήσουμε την απασχόληση αν δεν κάνουμε προσπάθεια σε όλες τις περιφέρειες. Πώς θα αυξηθεί το ποσοστό χρήσης των ανανεώσιμων ενεργειών αν δεν το κάνουμε σε όλες τις περιφέρειες. Και το ποσοστό έρευνας επομένως πρέπει να αυξηθεί σε όλες τις περιφέρειες ώστε να φτάσουμε στο 3% συνολικά στον ε, μέσον όρο της Ευρώπης. Άρα επιτυχής πολιτική και επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής θα γίνει μόνο με συμμετοχή των περιφερειών και επομένως η περιφερειακή πολιτική καλείται εδώ να αποδώσει. Επίσης, άλλο θέμα είναι ότι πρέπει ήδη από τώρα να αρχίσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής 2020 και στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Η ΔΕΜΗ θα τεθεί το θέμα πότε θα εφαρμοστεί η Ευρώπη του 2020. Αν περιμένουμε μέχρι το 2014 νομίζω ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Υπάρχει και υπολογισμός που έχει κάνει του κυρίου Λεβαντόφσκι που δείχνει ότι τα κονδύλια που ήδη τώρα διατίθενται στις περιφέρειες εξυπηρετούν κατά 60% τους στόχους στρατηγικής 2020. Αυτό οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε και τα επόμενα τρία χρόνια. Να αρχίσουν λοιπόν να εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα. Υπήρξε και μια αρκετά κριτική συζήτηση σχετικά με την αιρεσιμότητα. Ενδεχομένως, και δεν το αποκλείω, Ορισμένοι έχουν δυσκολευτεί με τον όρο αυτό. Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε ότι ο στόχος είναι εδώ στην αρχή μιας περίοδου να συμφωνήσουμε πάνω σε όρους που πρέπει να πληρούνται για να γίνει να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα στις διάφορες περιφέρειες με τρόπο διαρκή και βιώσιμο. Νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνήσουν ότι υπάρχουν πολλά πρακτικά παραδείγματα καθυστέρησης της εφαρμογής ή της υλοποίησης έργων και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τόσο τα χρήματα που λείπουν, είναι περισσότερο ζητήματα ικανοτήτων, γνώσεων, πείρας ενδεχομένως μη διαθεσιμότητα των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων, μη ε, ικανοποιητικής εφαρμογής ευρωπαϊκών διατάξεων και μεταφοράς τους στα εθνικά δίκαια. Αυτά όλα είναι γνωστές συνθήκες που ισχύουν σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω μετά από τις σχετικές συζητήσεις κατανόησαν οι αρμόδιοι υπουργοί ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι κάτι που τους βοηθεί και τους ίδιους στην καθημερινή τους εργασία επιτόπου. Αν δηλαδή εδώ λαμβάνονται κάποιε αποφάσει οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται μετά ώστε να μπορούν να προχωρούν γρηγορότερα τα έργα. Έγιναν συζητήσει επίση για το αποτελεσματικό απόδοση για το, συγγνώμη, το αποθεματικό απόδοσης που δεν θα ανακατανέμεται ευρωπαϊκά αλλά το πολύ εθνικά. Δηλαδή θα υπάρχει ένα είδος ανταμοιβή ενδοκρατικής. Κατά την αντίληψη τη δική μας χρειάζεται τήρηση περίπου ενός περιθωρίου 2% του προϋπολογισμού θα προχωρήσουμε και σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση θα γίνει στη βάση αυτής ανακατανομή στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών και τη συνθήκη βρίσκονται πέραν των στόχων. Τι εννοώ δηλαδή. Είναι σημαντικό όταν εκφράζεται η ανησυχία αιτιολογημένη ή μη αιτιολογημένη τέλο πάντων αυτό ανεξαρτήτως. Αλλά διατυπώνεται η ανησυχία ότι το λεγόμενο performance reserve είναι κάτι το οποίο πηγαίνει μονάχα στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό στόχο. Αυτό είναι λάθος οι ευρωπαϊκοί στόχοι είναι κοινοί στόχοι που αποτελούν λίγο πολύ μια μέση τιμή. Και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν όλες οι περιφέρειες. Παράδειγμα, ανανεώσιμες ενέργειες. Ήδη σήμερα έχουμε περιφέρειες που, έχουν ήδη, που πληρούν ήδη το 20%. Θα ήταν λάθος να πούν τώρα σταματάμε, έχουμε φτάσει το 20%, ας κάνουν την προσπάθεια οι υπόλοιποι. Πρέπει να παραμείνουν στην προσπάθεια και να βάλουν νέους κατάλληλους στόχους, ας πούμε 40%. Και εάν αποδειχθεί σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση ότι μπορούν ίσως να φτάσουν και το 40% και το 45% τότε αυτή η περιφέρεια είναι υποψήφια για ε, την πρόθεση αυτή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει όμως και για μια περιφέρεια η οποία για παράδειγμα έχει φτάσει στο 10% δηλαδή το μισό του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Για την περιφέρεια αυτή όμως μπορεί να είναι φιλόδοξος ο στόχος και ίσως να δούμε τότε ότι μπορεί να φτάσει όχι μόνο το 10 αλλά και το 12-13%. Επομένως και αυτή μπαίνει τότε ε, υποψήφια για αυτό το performance reserve, το αποθεματικό απόδοσης. Πριν τώρα έλθω στο χρονοδιάγραμμα, να σας πω λίγα λόγια για τον προϋπολογισμό. Ειδικά εδώ, ενώπιόν σας, αλλά και στο Κοινοβούλιο συνολικότερα, έχω την αίσθηση ότι στην βάση των κοινών επιτευγμάτων μας τους τελευταίους μήνες που εκδηλώνονται και στην δημοσιονομική ενδιάμεση έκθεση όπου η περιφερειακή πολιτική επανακτά έδαφος και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον προϋπολογισμό και την θέσπιση του δεν έχει λήξει προσπάθεια διότι πρώτον τίθεται το ερώτημα ποια θα είναι η τελική μορφή του συνολικού προϋπολογισμού και αυτό λοιπόν θα συζητηθεί και μέσα σε αυτό το συνολικό προϋπολογισμό το τμήμα της περιφερειακής πολιτικής ποιο θα είναι. Άρα προσοχή. Μην θεωρήσουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλείς και μπορούμε να επαναπαθούμε και ότι έχει λήξει η προσπάθειά μας. Θα έλεγα μάλλον την έχουμε βγάλει ας πούμε από το ψυγείο. Αυτό είναι. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ας συνεχίσουν να επαγρυπνούν και ας φροντίζουν και φροντίζουμε όλοι ώστε να εξασφαλιστεί ότι και στο μέλλον σε απόλυτους αριθμούς θα έχουμε στα χέρια μας ένα λογικό προϋπολογισμό που να βρίσκεται περίπου σε τάξεις μεγέθους του σημερινού, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τα έργα τα οποία μας απασχολούν. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές εκείνους που ήδη με εκθέσεις και ούτω καθεξής παρακολουθούν τις εξελίξεις φροντίζουν έτσι ώστε να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση. Δεύτερο σημείο τώρα για τον προπολογισμό εξακολουθούν οι συζητήσεις σχετικά με τη διάρκεια της ε, δημοσιονομικής περίοδου. Ακούω κάποιους να μιλούν για πέντε χρόνια, ταυτόχρονα όμως θεωρούν ότι η περιφερειακή πολιτική λόγω πολιετούς χαρακτήρα χρειάζεται 7 χρόνια. Νομίζω από τη δική μας σκοπιά, ή τουλάχιστον τη δική μου σκοπιά, δεν το κρύβω, ε, είναι λογικό χρονικό διάστημα. Υπάρχει και η πρόταση Μπαρόσο, εξακολουθεί και υπάρχει η πρόταση Μπαρόσο, 5 συν 5. Αλλά εν τέλει νομίζω ότι μόνο 5 χρόνια από τη σκοπιά της περιφερειακής πολιτικής αποτελούν στην ουσία δύσκολο εγχείρημα. Γιατί πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν οι πολιτικές αυτές. Είναι η φάση roll-out πρώτα. Για του χρόνου έχουμε ξεκινήσει μεγάλη διαδικασία διαβουλεύσεων Ιανουάριο και αρχές Φεβρουαρίου στο λεγόμενο Cohesion Forum, το βήμα συνοχής, με συνεισφορές, συμβολές, συμβολές θα δοθεί, θα γίνει νέα έκθεση που θα αποτελέσει πλέον την βάση για τις νέες μας εργασίες για να υποβάλουμε τα νέα σχέδια κανονισμών περί τα μέσα του έτους και λίγο πολύ ταυτόχρονα με την πρόταση για την μελλοντική δημοσιονομική περίοδο. Αυτά συνδέονται τα πράγματα και περί τα τέλη του έτους, κύριε Πρόεδρε, θα υποβάλουμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο διαφόρων ταμείων, γεωργίας, αλίας, διαρθωτικά ταμεία για να βολιδοσκοπήσουμε, να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να βελτιωθεί η απόδοση επιτόπου. Αυτά είναι τα θέματα επί των οποίων ήθελα ιδίω να εφιστήσω την προσοχή σας. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω και με διάφορες πολιτικές ομάδες για τα διάφορα θέματα. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Τα όσα σας είπα αποτελούν μια απήχηση λίγο της συζητήσεως που έχει διεξαχθεί από την λήψη της αποφάσεως πριν από ένα μήνα περίπου και των διαφόρων πτυχών που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτήν τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και θα ήθελα να αρχίσω με τον κύριο Φανίστερο σας παρακαλώ συνάδελφοι γενικά να μην επεκτείνεστε διότι έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Με ναι, Λάμπερ, έχεις το λόγο. Θα ήθελα να θίξω τρία σημεία, κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα μία απάντηση σε αυτά τα σημεία. Αν λάβουμε υπόψη την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην, στις εργασίες μας, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο Επίτροπος μπορεί να μας διευκρινίσει το πώς έχουν οι κανονισμοί. Θα υπάρξει ένας γενικός κανονισμός, ένας κανονισμός πλαίσιο και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρξουν ξεχωριστοί κανονισμοί για το ΕΤΠΑ και για τα ταμεία συνοχής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια να ξέρουμε ποια θα είναι η νομοθετική μας εργασία. Μερικοί λένε ότι θα χειριστούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Δηλαδή δεν θα έχουμε τρεις διαφορετικούς κανονισμούς, αλλά θα έχουμε μία ομαδοποίηση κανονισμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εργασία μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις συμφωνίες σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. Επίσης θα ήθελα να τονίσω το εξής. Όταν διαβάζω σελίδα 18 του ανακεφαλαιωτικού αυτού εγγράφου μιλάτε για τη συνεισφορά των κρατών μελών σε σχέση με εταιρικέ σχέσεις, συμβάσεις και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς οι δεσμεύσεις αυτές οδηγούν σε ένα κοινό πλαίσιο μεταξύ κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο ρόλο θα διαδραματίσουν οι πόλεις και οι περιφέρειες, γιατί μιλήσαμε για μία περιφερειακή ε, σύμβαση η οποία θα πρέπει να υπογραφεί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους όρους που έχει θέσει η Επιτροπή. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ποιες είναι οι δεσμεύσεις των κρατών μελών για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δεν αρκεί να έχουμε στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, ε, πληροφορίες για το πόσο θα υπάρξει μια περιφερειακή καθαρά σύμβαση. Μιλήσατε για 7 χρόνια ή 5 συν 5. Πολλές φορές όμως χρειαζόμαστε ένα δεκαετές πλαίσιο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγματα επ' αυτού. Μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα 5 συν 5 με ειδική θέση για τα καινοτόμα σχέδια για συγκεκριμένα διαρθρωτικά σχέδια ως προς ε, επιστημονικά σχέδια και ερευνητικά σχέδια. Αυτές είναι οι τρεις μου ερωτήσεις. και πιστεύω ότι τα καταφέρατε πολύ καλά. Äh, äh, Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε από την περίοδο χρηματοδότησης. Στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα τη συζήτηση και στην πραγματικότητα μιλάμε για την ομοθεσία του Κοινοβουλίου καθαρά. έτσι ώστε να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση και την ιεράρχησή της. Έγινε λόγος για πέντε χρόνια και για την ΚΑΠ και για την διαρθρωτική πολιτική. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε έμπρακτα πώς θα λειτουργούσε αυτό το ε, πλαίσιο. Θα έχουμε έναν δημοσιονομικό προγραμματισμό δύο τρίτων για 5-7 χρόνια και 1 τρίτον για 5 7 χρονια και 1 τριτων για 5 χρονια Θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Επίσης ακούστηκαν φήμες ότι η Κομισιόν θα υποβάλει μία κοινή πρόταση για τα εν λόγω ταμεία και το περιφερειακό ταμείο. Εμείς είχαμε αντιταχθεί σε κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ίσως μπορεί να μας το διευκρινίσει ο Επίτροπος Πρόεδρε. Ως προς την αιρεσιμότητα για τα κράτη-μέλη, θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση και σε αυτόν το τομέα γιατί υπάρχει πολλαπλή ερμηνεία της αιρεσιμότητας. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο γίνεται μία διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη ως προς τις προτεραιότητες. Δηλαδή, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κοινής απόφασης. Μιλάμε για την Εθνική Ένωμη Τάξη και ε, εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το ζήτημα, διότι θα πρέπει να βρούμε ένα μέσον οικονομικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Ε, διάβασα το έγγραφο και έχω ορισμένες ερωτήσεις. Βεβαίως, Υπάρχουν ήδη σχέδια που μιλούν για αιρεσιμότητα και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα αιρεσιμότητας που σχετίζονται με πολιτικούς στόχους συνοχής. Στο έγγραφο είδα ότι έχουν εισαχθεί μέτρα αιρεσιμότητας που δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική συνοχή Σε περίπτωση παραβίασης του Συμφώνου ε, Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε πώς θα κινηθούμε προς την πρόοδο των σχεδίων, αλλά θα υπάρχουν και κυρώσεις έναντι των κρατών μελών με βάση την πολιτική συνοχής. Δηλαδή θα αλλάξουμε την πολιτική συνοχής ε, και θα την ε, οδηγήσουμε σε μία διαχείριση, μία διορθωτική διαχείριση προς τα κράτη-μέλη. Γιατί όπως ξέρετε και σε προηγούμενες συναντήσεις είπαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μία καθαρά κυρωτική πολιτική. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τις ε, τοπικές αρχές και τους δικαιούχους και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αντίθετο πλαίσιο, δηλαδή να προβούμε σε κυρώσεις κατά των κρατών μελών. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι σωστό εξαιτίας των κυβερνητικών σφαλμάτων να υποστούν κυρώσεις οι δικαιούχοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εφαρμόζονται σωστά τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα ήθελα από αυτού του θέματος να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις. Επίσης, η Επιτροπή προβλέπει αυστηρά μέτρα σε σχέση με την διαχείριση των προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχει ένας ετήσιος απολογισμός με βάση τις ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί για την πολιτική συνοχή. Τι κάνουμε όμως για τα πολιετή προγράμματα. Βεβαίως αυτά τα σχέδια μπορούν να ισχύσουν για την ΚΑΠ. Στην περίπτωση των Ταμείων Συνοχής έχουμε και πολιετή προγράμματα και εδώ ίσως ανακύψουν τεχνικά προβλήματα τα οποία στην ουσία οδηγήσουν σε επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Δηλαδή να υπάρχει ένας υπερέλεγχος τον οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε μια ενιαία διαδικασία ελέγχου και διάλογο με τις τοπικές αρχές. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, συνεπείς, έτσι ώστε αυτά τα μέτρα να αντικατοπτρίζουν μία πραγματικότητα. Δηλαδή τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφέρθω αφορούν την βελτίωση της απόδοσης των κρατών μελών. Πώς θα το ελέγξει αυτό η Κομισιόν, γιατί πρόκειται για ένα περίπλοκο σχέδιο και από το κείμενο δεν είναι σαφές πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση και πώς θα ε, εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε ε, να ευεργετηθούν οι δικαιούχοι μακροπρόθεσμα και να μην υπάρχουν προβλήματα ως προς τις επιστροφές εξόδων στις αγορές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε έναν επιπρόσθετο, ε, ένα επιπρόσθετο άχθος από πλευράς γραφειοκρατίας. Επίσης πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε πραγματικά την κατάσταση ως προς την πολιτική συνοχής. Τους τελευταίους μήνες είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία και προτείναμε μέτρα προς την Κομισιόν. Δηλαδή, πέρα από θέματα αρχής, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προσυγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των δικαιούχων. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ για αυτές τις ε, διευκρινήσεις που μας κάνατε ως προσορισμένα θέματα της πρότασης της πρότασης της Επιτροπής, αυτής της πέμπτης έκθεσης για τα Ταμεία Συνοχής. Ωστόσο, μένουν μερικά θέματα ανοιχτά. Είπατε ότι θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενισχύσεις όλες οι ε, περιφέρειες ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν και να επιτύχουν τους στόχους του 2020. Πώς θα το συνδυάσετε αυτό με το γεγονός ότι τα χρήματα έχουν λιγοστεύσει. Ήδη αυτό είναι ένα γεγονός. Πώς θα το συνδυάσετε με το γεγονός ότι θέτει ε, στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής τη συνθήκη κυρίως στις πιο μειονεκτικέ περιοχές. Πώς θα το επιτύχετε λοιπόν αυτό. Εδώ ήσασταν λίγο ασαφεί. Όχι υποσχέσεις, πράγματα τα οποία που μπορούν, να, μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό θέλω να ακούσω. Δεύτερο, η συνθήκη ανάπτυξη. Όπως έχω ακούσει από τη Γενική σας Διευθύνση, είναι ένα είδο συνθήκης το οποίο θα καταστρώσει το στρατηγικό πλαίσιο και θα το κάνει δεσμευτικό. Δεν σημαίνει αυτό ότι προτιμάτε τότε το κυβερνητικό επίπεδο, το ανώτατο επίπεδο των κρατών δηλαδή και όχι η Ευρώπη των περιφερειών. Αυτό που δεν είναι καθόλου σαφές είναι που βρίσκεται η αρχή της συνεταιρικότητας. Οι εταίροι απλώς είναι θεατές, διότι στην ουσία πρόκειται για διακρατική συμφωνία ή τουλάχιστον για συμφωνία μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων. Και στο εγγραφό σας δεν λέτε τίποτε το νέο, δεν αναφέρεστε καθόλου σε αυτή τη ε, σχέση. Ήδη στην συνθήκη αυτή ασκείται πολύ έντονη κριτική, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών από τις κυβερνήσεις. Αλλά αφήνει απ' έξω την περιφερειακή πολιτική στην ουσία. Άλλωστε και εμείς επικρινόμαστε μαζικά για το λόγο αυτό. Και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και πολλά πράγματα σε αυτούς που μας επικρίνουν, διότι είναι πολύ νεφελώδη τα πράγματα. Βλάσακ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές και να τονίσω τον ρόλο της συναπόφασης και τις συζητήσεις για τους μελλοντικούς στόχους, αλλά επίσης να δούμε πώς μπορούμε να επανορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να γίνει μια σαφής ανάλυση των ε, μεμονωμένων σφαλμάτων και προσωπικά θα ήθελα να μου πείτε πώς έχει η κατάσταση. Δεν έχουμε διερμηνία προς τα γερμανικά. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω και θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι σημαντική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με βάση μια προσέγγιση εταιρικών οικονομικών σχέσεων. Αυτό αποτελεί εγγύηση για αποδοτικά αποτελέσματα όταν λοιπόν προετοιμάζουμε ε, νέα προγράμματα θα πρέπει να δούμε αυτές τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις και να υπάρχει χνηλασιμότητα όλων των σφαλμάτων. Θα ήθελα να επενέσω την εργασία της ε, Επιτροπής, ιδιαίτερα στο θέμα της ε, αστικής συνεργασίας, της εδαφικής συνεργασίας, ιδιαίτερα ως προς τις ε, κομοπόλεις, τις αγροτικές περιοχές και τις μεγαλουπόλεις. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία στενή συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των χωροταξικών δομών. Πώς θα το εγγυηθείτε αυτό. Θα θέλαμε να μας απαντήσει η Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω λίγο ερωτήσεις που έκαναν επί διαφόρων θεμάτων οι συντονιστές για το θέμα της συναπόφασης. Προσπαθώ και σε πολλές εκδηλώσεις ή διοργανώσεις που επισκέπτομαι και στις χώρες μέλη προσπαθώ να δημιουργήσω την συνείδηση ότι ιδίω η διαμόρφωση του προγραμματισμού και οι διαπραγματεύσεις για τον προγραμματισμό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μοναχά ανάμεσα στην Κομισιόν και στις χώρες μέλη αλλά ότι πρέπει να εντάσσονται στην προσπάθεια και οι περιφέρειες. Και όχι μόνο οι περιφέρειες, αλλά και το τοπικό επίπεδο, διότι διαπιστώνω σε τέτοιες συναντήσεις ότι το τοπικό επίπεδο παραπονείται ήδη ότι τα πράγματα μένουν στο περιφερειακό, στο επίπεδο της περιφέρειας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά φίλτρα όπου τα πράγματα μπορούν να κολλήσουν. Πρέπει όλες, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να συμμετέχουν γιατί μόνο τότε γίνεται και αυτή η ταυτοποίηση του πολίτη και του επίπεδου με την απόφαση. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι βέβαια να βγω από τα θεσμικά πλαίσια. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επισημαίνω να βλέπω βέβαια και ποιος συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις το μόνο που μπορώ να κάνω είναι επιμένω να επισημαίνω την ανάγκη ότι πρέπει να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα. Κυρία Σρόιντερ, απαντώ σε εσά. Η συνθήκη εταιρικότητας και επενδύσεων είναι διαμορφωμένη και στα πλαίσια ή θα πρέπει να διαμορφωθεί και να συναρθεί και στα πλαίσια των θεσμικών περιορισμών. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου ως γνωστόν τα ομόσπονδα κρατήδια της έχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση μέσα στην δομή του κράτους αυτού. Υποθέτω ότι σε τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, σε τέτοιο συνταγματικό πλαίσιο, θα χρειαστεί μια συμφωνία που θα περιορίζεται να καλύπτει εθνικά θέματα. Έχουμε εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο, για παράδειγμα, για τη Γερμανία στο τομέα των μεταφορών. Εκεί να υπάρξουν και επιχειρησιακά προγράμματα που να εγκριθούν και στο επίπεδο των ομόσπονδων κρατηδίων. Ακόμα δεν έχουμε αποκρεσταλώσει άποψη. Όπως όμως εξελίσσεται μέχρι τώρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε ειδικά ανά κράτος σε ό,τι αφορά τον τύπο. Σε ό,τι αφορά την ουσία, εμείς θα κάνουμε προσπάθεια ώστε στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις να συμμετάσχουν κατά το δυνατόν όλα τα επίπεδα. Εδώ πάλι με την ευκαιρία θα πω ότι εμείς κάνουμε και διαφήμιση των εισαγωγικών, προωθούμε την ιδέα δηλαδή ότι πρέπει να μην μείνει το πράγμα, να μην κολλήσει το πράγμα στο επίπεδο της περιφέρειας, αλλά πρέπει να συμμετάσχει και το τοπικό επίπεδο. Για το θέμα των κανόνων και κατά πόσο θα ενοποιηθούν. Έχουμε να λάβουμε υπόψη και το συμφέρον των χρηστών να υπάρχουν ή δυνατόν ενιαίοι κανόνες και ιδίω, αλλά αυτό βέβαια συζητείται ακόμα μεταξύ EADF και ESF ώστε και αυτή είναι τουλάχιστον δική μου προσέγγιση να υπάρχουν για τα δύο αυτά τα μία τελικά ορισμένοι ειδικοί κανόνες αλλά να μην υπάρχει από την αρχή ο μέγιστος δυνατός διαχωρισμός. Στόχος είναι να υπάρχει μια λίγο πολύ κοινή προσέγγιση και για το Ταμείο Συνοχής το εξετάζουμε αυτό γιατί και πέρα και από το γεγονός ότι το Ταμείο έχει κάπως περιορισμένη ε, ικανότητα ενισχύσεως για ορισμένους τομείς. Για ορισμένες περιφέρειες χρήματα αντλούνται από διάφορα ταμεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ακούω διάφορες αξιώσεις, διάφορες απαιτήσεις για να υπάρξει μια εναρμόνιση. Βέβαια, ορισμένες ιδιαιτερότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για τους όρους, για την αιρεσιμότητα τώρα, επανέρχομαι, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι γίνεται μια συζήτηση η οποία ξεφεύγει και από τα όρια της περιφερειακής πολιτικής. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε χώρες μέλη από το ευρωπαϊκό επίπεδο που κατ' επανάληψη έχουν παραβιάσει συμφωνίες όπως για παράδειγμα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξο άνθρωπος και έχω την ελπίδα ότι μια ακαδημαϊκή συζήτηση και με τις χώρε αυτέ οι οποίες έχουν κατ' επανάληψη παραβιάσει τις συμφωνίες αυτές θα επιτρέψει να αποκαταστήσουμε πάλι το πλαίσιο και την προσπάθεια αυτή. Έχουν συζητηθεί, έχει συζητηθεί μάλλον και το ενδεχόμενο κυρώσεων. Ορισμένοι νομομαθείς διαπιστώνουν ότι ήδη σήμερα στους κανόνες του Ταμείου Συνοχής υπάρχει κάποια παράγραφος που θα μπορούσε να βασίσει την αναστολή κάποιων υπεσχημένων. Αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ αυτό. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορισμένοι συνάδελφοι και όχι λίγοι, έχουν διαπιστώσει ότι αυτό ο μηχανισμό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ούτω ή άλλω διότι θα έπλητε μόνο 15 χώρε και όχι τι υπόλοιπε 12. Το θέμα λοιπόν των κυρώσεων, στο θέμα των κυρώσεων μάλλον, έχει, έχουμε καταλήξει στην σκέψη ότι αν υπάρξουν κυρώσει, θα πρέπει να τίθεται επιτάπητο ολόκληρο ο κοινοτικό προπολογισμό μια χώρα. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση. Ο συνολικό κοινοτικό προπολογισμό και αυτό βεβαίως έχει σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Στην έκθεση συνοχής και στα συμπεράσματα στα συμπεράσματά της θα πρέπει να περιληφθούν ωστόσο στοιχεία που αναφέρονται σε ολόκληρο τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, τα χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων έχουν το νόημα, ειδικά σε δύσκολου καιρού, να δώσουν κάποια νέα πνοή στην οικονομία. Επομένως, μια τέτοια προσέγγιση θα είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Επιβολή κυρώσεων δηλαδή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αποφευθεί εφόσον είναι δυνατόν. Και στο άτυπο ε, Συμβούλιο Υπουργών έγιναν διεξοδικότατες συζητήσεις από ό,τι διαβάζω στα πορίσματά τους όπου γενικά ο τόνος των συζητήσεων ήταν ότι δεν γίνονται αποδεκτές μακροοικονομικές αιρεσιμότητες. Και οι παρόντες υπουργοί δεν δέχονταν αιρεσιμότητα που να αναφέρεται στην πολιτική συνοχής. Και αυτό για μένα είναι και το σημαντικότερο. Διότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον να εφαρμοστούν τα έργα, να υλοποιηθούν τα έργα. Σε ό,τι αφορά τα auditing τώρα, τους δημοσιονομικούς ελέγχους, είπα ήδη ότι πρέπει να δούμε ότι οι χώρες μέλη βάζουν και άλλους κύκλους ελέγχων, είναι υποχρωμένες και εκ του συστήματος. Μπορούν βέβαια να απροποιηθούν ορισμένα πράγματα, και να εναρμονιστούν, αλλά ας μην λησμονούμε ότι και πάλι εδώ υπάρχουν ειδικέ νομοθεσίες των χωρών μελών που επίσης την χάνουν εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά την οικονομική τώρα διάσταση, κυρία Σρέντερ, έχω πει ξανά ότι χρειαζόμαστε έναν λογικό προϋπολογισμό και από τη σκοπιά μου αυτό σημαίνει ότι σε απόλυτους αριθμούς θα πρέπει να είναι περίπου όπως ο σημερινός, ο τωρινός. Εάν ο μελλοντικός προϋπολογισμός σε απόλυτους αριθμούς απέχει σημαντικά από τον τωρινό, ορισμένα πράγματα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έχουμε ήδη περιφέρειες που λόγω μεγέθους, δηλαδή σχετικά μικρού μεγέθους ή έχουν λίγο κόσμο, δεν παίρνουν πολλά χρήματα. Εάν εδώ πέσουμε κάτω από μια ορισμένη τάξη μεγέθους, δεν θα μπορούμε ούτε πλέον να αντιμετωπίζουμε το διοικητικό κόστος του προγράμματος. Δεν θα μπορούσα να σας πω πού βρίσκεται αυτό το ελάχιστο όριο, αλλά εγώ πάντως θεωρώ σημαντικό ένα προϋπολογισμό σε απόλυτους αριθμούς και όχι σε ποσοστά. Σημαντικό να είναι λοιπόν στα επίπεδα τα σημερινά. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την σχέση μεταξύ περιφερειών συγκλήσεως και περιφερειών ανταγωνισμού που είναι περίπου στο 1 προς 10 η αναλογία αυτή, αν μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον και με την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ θα ήθελα να σας πω ότι και κυρίως απευθυνόμενος στους βουλευτές χωρών απολυπτριών, να το πω έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δική μου, κατά τη δική μου πολιτική κρίση, εφόσον υπάρξει μειωμένος προϋπολογισμός, ίσως προκύψει μια κατάσταση όπου τα χρήματα πλέον των θα ταμείων θα πάνε μοναχά στις περιφέρειες συνοχής και τότε οι εύπορες ας πούμε χώρες δεν θα λαμβάνουν τίποτα. Στις χώρες καθαρούς εισφορείς, για παράδειγμα Γερμανία, έχουμε ξεκάθαρες αποφάσεις για να περάσουν χρήματα του Περιφερειακού Ταμείου στις ε, περιφέρειες ανταγωνισμού. Εάν τώρα μειωθούν τα χρήματα του Περιφερειακού Ταμείου, θα αντιμετωπίσουμε ποσοστιαίες μειώσεις, αναλογικές μειώσεις. Και αυτό βέβαια θα πλήξει τους beneficiaries, τους απολύπτες των χρημάτων αυτών. Πέραν του ότι αυτό που είπα πριν για την εφαρμογή της στρατηγικής 2020 δεν πρόκειται να λειτουργήσει βέβαια με τέτοιο τρόπο. Και εδώ έχουμε 84 περιφέρειες που είναι περιφέρειες σύγκλησης και όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θεωρώ ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα έχουμε κάτω από 70 περιφέρειες θα δούμε και τον αριθμό πληθυσμού σε περιφέρειες συγκλήσεως έχουμε μέχρι τώρα 155 εκατομμύρια κατοίκους εάν συνεχίσουν να εξελίσσονται οι αριθμοί όπως το βλέπουμε τώρα, στην επόμενη, στην επόμενη περίοδο θα έχουμε μόνο 120 εκατομμύρια άτομα που κατοικούν σε περιφέρειες συγκλήσεως. Κάτι το οποίο αφενός δείχνει την επιτυχία κάπως πιο μακροπρόθεσμα της πολιτικής αυτής, δείχνει όμως ταυτόχρονα ότι απελευθερώνονται και κάποια κονδύλια που μπορούν να δοθούν αλλού, ώστε στο σύνολο να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες και πράγματι, με ένα, όπως είπα, λογικό προϋπολογισμό, όλες οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τώρα η άλλη δική σας ερώτηση ήταν για την διασύνδεση με την απόδοση. Αυτό εξαρτάται από το ποσοστό ή από τους απόλυτους αριθμούς. Αυτό θα το δείξουν οι συζητήσεις των επομένων εβδομάδων και μηνών. Δηλαδή, πρώτον, εάν το έργο αυτό πραγματικά, α, το project αυτό θα επιβιώσει, κάτι που ελπίζω, και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η ανακατανομή. Θα χρειαστεί μια συνολική ευρωπαϊκή ανακατανομή, κατά τη γνώμη μου, ώστε τα κονδύλια να κατανεμηθούν στις περιφέρειες Για την ώρα πάντως θεωρώ πρόημο να, να δώσω μια απάντηση πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Μας μένουν 10 λεπτά και 11 αγορητές. Διότι ο Επίτροπος θέλει να μας παρουσιάσει και τη στατική του Δούναβη για την οποία θα μας μείνουν 10-15 λεπτά. Έχουμε όπως είπα λοιπόν ένα δεκάλεπτο 11 αγορητές Ακόμα και αν φανείτε πάρα πολύ πειθαρχική και μιλήσετε για λιγότερο από ένα λεπτό, πάλι δεν προλαβαίνουμε. Άρα η πρόταση είναι να Έχετε το λόγο. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Διότι στην ε, επεξήγηση της Κομισιόν είχαμε την ε, την ε, παρουσίαση της έβδομης έκθεσης συνοχής και νομίζω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να βρούμε νέο χρόνο, διότι έλαβα απαντήσεις έτσι, αλλά θα πρέπει να έχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορώ να δω πώς θα διαχειριστούμε τον κανονισμό, πώς θα προετοιμαστεί δηλαδή. Σας ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δεν μας απαντήσατε επακριβώς. Θα ήθελα να βρούμε χρόνο για να μπορούμε να συζητήσουμε με την Επιτροπή πριν από το Φόρουμ Συνοχής. Ο Επίτροπος θα επανέλθει τον Ιανουάριο επί του θέματος. Νομίζω ότι πέντε πρέπει να λάβουν το λόγο, αλλά η παρέμβασή σας να είναι κάτω του ενός λεπτού. Θα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά οι επόμενοι θα λάβουν το λόγο των Ιανουάριο. Η κυρία Ιριγκόιαν που είναι νέο μέλος από όσο καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα κοιτάξω να είμαι πολύ σύντομη. Και σύντομα θα ρωτήσω. Τηρώντας το ένα λεπτό. Για τις διαρθρωτικές πολιτικές η χρηματοδότηση ολοκληρώνεται σε περιφερειακή κλίμακα. Χρειάζεται λοιπόν πάντα να έχουμε στρατηγικές ενεργητικής ανάπτυξης, δηλαδή και φυσικούς αλλά και άειλους πόρους. Τι σκέφτεται γι' αυτά η Κομισιόν για να μπορέσει να ενισχύσει το αναπτυξιακό επίπεδο. Για το θέμα τώρα της δημογραφίας και της απερίμωσης από τον πληθυσμό τους των ε, απομονωμένων και νησιωτικών περιοχών. Η Καστίγια Ηλεών που είναι η εκλογική μου περιφέρεια υποφέρει από αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ε, για την πρόκληση της γύρανσης του πληθυσμού, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν στα πλαίσια της μελλοντικής πολιτικής συνοχής ούτω ώστε να λάβει υπόψη τη την, ε, ε, ε, τη γύρανση του πληθυσμού και την δημογραφική μείωση. Για τους στόχους τώρα σύγκλησης, στην πέμπτη έκθεση αναφέρεται να δημιουργηθεί μία ενδιάμεση κατηγορία των περιφερειών που θα αντικαθιστούσε το facing out και το facing in θα μπορούσε να μας πει λοιπόν ο Επίτροπος ε, τι ε, σκοπεύει να κάνει το μέσο των ε, μεταβατικών περιόδων για τη βοήθεια τι ρόλο θα έχει στη νέα αυτή πολιτική ένα λεπτό και μία ερώτηση σας παρακαλώ συνάδελφοι πρέπει να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ο κ. Στραμόπουλος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Δύο σημεία. Πρώτον, πολύ σύντομα, πώς εκτιμά ο κ. Επίτροπος το ότι και πώς ακριβώς θα επηρεάσει η κρίση, η δημοσιονομική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα κάποιε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, πώς θα ε, επηρεάσει τις ε, χρηματοδοτήσεις με δεδομένο ότι ακούμε απόψεις ότι οι χώρες που έχουν δημοσιονομικά, δημοσιονομικά προβλήματα θα πρέπει και να τιμωρηθούν κατά κάποιο τρόπο και όσον αφορά την ε, περιφερειακή πολιτική. Και δεύτερον, εδώ στην ε, Επιτροπή υιοθετήσαμε και μετά στη συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο την, ε, μια έκθεση με προτάσεις για τη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές περιφερειακές χρηματοδοτήσεις. Την έχετε πάρει υπόψη στις πολιτικές και πώς εκφράζεται αυτό.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 Έχω πάρα πολλά θέματα να αναφέρω. Θα σταθώ όμως σε ένα μόνο, αστική πολιτική. Ξέρετε ότι είναι κάτι το ουσιαστικό για μένα ε, μέσα στην μελλοντική πολιτική συνοχή ως αντιπρόεδρος του Ουρμπαν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Και δεν είναι κάτι το οποίο αντιπαρατίθεται στην πολιτική για την Ήπεθρο. Είναι δύο συμπληρωματικές πολιτικές. Με ανησυχεί όμως κάτι η πολιτική για την Ήπεθρο. Στην πέμπτη έκθεση για τη συνοχή δεν αναφέρεται σχεδόν και σε όλα τα έγγραφα τα οποία συζητιούνται και παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο, Στρατηγική 2020 κτλ. δεν εξετάζουν ε, επαρκώς την ε, διάσταση της υπαίθρου. Πολλές φορές αποσιάζει εντελώς απολυσμένα έγγραφα θα ήθελα να με διασφαλίσετε για αυτό το θέμα και να μου πείτε ότι στο μέλλον θα έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΦΕΝΤΕΡ και ΦΕΑΝΤΕΡ και δεν θα πρέπει να ε, αγνοήσουμε την χωροταξική συνοχή μέσα στα πλαίσια όλων των πολιτικών και διαστάσεων της περιφερειακής πολιτικής. Μισό λεπτό ο Μίχαλ Τόιρερ. Is Mikael with us? No, he's not. That... Α, δεν είναι παρόν ο Μίχαλ. Καλά. Τότε παρακαλώ κύριε Επίτροπε, απαντήστε. Okay. Καλά λοιπόν, σχέδιο ανάπτυξης. Είναι σημαντικό οι περιφέρειες να αρχίσουν από τώρα να προπαρασκευάζονται για τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το 2013. Υπάρχει ένας αριθμός ανακοινώσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για την διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδίου. Πρόκειται για συζητήσεις που πρέπει να διεξαγάγουμε με τις περιφέρειες, με το τοπικό επίπεδο και με τις χώρες μέλη. Αλλά βέβαια είναι και προτάσεις, πρέπει να γίνουν μάλλον και προτάσεις από τις περιφέρειες και από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει και για τι 273 περιφέρειες τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Όπως το βλέπουμε εμείς, εμείς είμαστε εδώ ως συνομιλητές, είμαστε διαθέσιμοι ως συνομιλητέ ως μέτοχοι στι διαπραγματεύσει για τους στόχους που πρέπει να είναι φιλόδοξοι, στόχοι αλλά και ρεαλιστικοί. Να δούμε αν τα, αν τα προγράμματα βρίσκονται σε συμφωνία με ε, τη στατική του 2020. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση, αυτό είναι το δικό μας μέρος ε, της προσπάθειας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί η κάθε περιφέρεια, βεβαίως και εμείς έχουμε κάποιες ιδέες, αλλά πρέπει κυρίως να προέλθουν προτάσεις αυτές από τις ίδιες τις περιφέρειες. Και σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες μειονεκτικές ε, περιφέρειες δύσκολα προσβάσιμες κλπ. Το θέμα το δημογραφικό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο μας συνοδεύει διαρκώς. Δεν έχω απλές απαντήσεις όπως και κανένας δεν έχει. Παρακολουθώντας το φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη βλέπουμε μια απογύμνωση από κόσμο της υπαίθρου, μια φυγή προς τις πόλεις, προς τα αστικά κέντρα και νομίζω ότι κανένας από, κανένας δεν θέλει να συνεχίζεται το φαινόμενο αυτό. Η δική μου προσπάθεια είναι να συνεργαστούμε ή δυνατόν με κάθε μια περιφέρεια. Έχω ήδη επισκεφθεί πολλές περιφέρειες και τέτοιες που γεωγραφικά πραγματικά είναι μειονεκτικές. Και είναι, υπάρχουν αρκετές οι οποίες κατάφεραν να δώσουν και για τους εαυτούς τους, ας το πω έτσι, μια οικονομική διάσταση στην προσπάθεια αυτή, μια οικονομική διάσταση φτιάχνοντας αυτά τα ε, κέντρα διασποράς του, της ε, οικονομικής ανάπτυξης. Παράδειγμα, η προσπάθεια να υπάρξει εκπαίδευση, οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν επιτόπου εφόσον βλέπουν ότι έχουν κάποια δυνατότητα ανάπτυξης. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν αποδίδουν πρόθεσμα Είναι όμως πράγματα τα οποία αξίζουν να γίνουν και όπως είπα και, και οι περιφέρειες πρέπει να αρχίσουν ήδη την προσπάθεια. Ε, έχω πει για την σχέση μεταξύ αστικού κέντρου και υπαίθρου έχουμε δώσει ε, και ιδιαίτερη έμφαση και στο αστικό κέντρο, όχι μόνο διότι οι Ευρωπαίοι κατά 70% ζουν σε αστικά κέντρα, αλλά και διότι είδαμε και μέσα στην περίοδο προγραμματισμού ότι οι πόλεις, τα αστικά κέντρα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν είχαν λάβει αρκετά, ενώ ο χώρος της υπαίθρου έχοντας ιδιαίτερα προγράμματα, ιδίω για τον γεωργικό τομέα, αλλά και με τα δικά μας τα προγράμματα της περιφερειακής ανάπτυξης, είχαν μέχρι τώρα απολαύσει μια προτεραιότητα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την προσπάθεια σε εκείνα τα σημεία τομής ανάμεσα στο αστικό κέντρο και στην περιφέρεια και στην ε, Ήπεθρο και το Ταμείο της ανάπτυξης της υπαίθρου προσφέρει κονδύλια για το σύνολο της ανάπτυξης της υπαίθρου και όχι μόναχα για γεωργικές εκμεταλλεύσεις διότι στην Ήπεθρο υπάρχουν και άλλου είδους επιχειρήσεις εκτός από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ώστε λοιπόν η προσπάθεια πρέπει να, περιλάβει ολόκληρο τον χώρο της Υπέθρου δεν πρόκειται για καμιά, κανένας είδους αντίθεση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τονισμό που δίνεται επειδή έχουμε κατανοήσει ότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί κάποια ελλείμματα. Ξαναλέω, δεν τίθεται θέμα για την ώρα στις συζητήσεις επιβολής κυρώσεων και κυρίως για θέματα κονδυλίων των διαρθωτικών ταμείων. Οι συνέπειες λοιπόν της οικονομικής κρίσης εμφανίζονται και με το ότι ο ιδιωτικός τομέας σε πολλές χώρες διστάζει πολύ να επενδύσει και κυρίως όπου πρόκειται για πολυετή έργα, δηλαδή έργα πολυετούς προγραμματισμού. Εδώ βλέπουμε ακόμα, όπως είπα, δισταγμό, επιφύλαξη. Το, ο δημόσιος τομέας επενδύει περισσότερο, εν προκειμένου, και σε ό,τι μας αφορά με προκαταβολές ήδη το 2009 και 2010. Έχουμε προσφέρει επιπροσθέτως 7 δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες μέλη για να δώσουμε μεγαλύτερη ρευστότητα προς την κατεύθυνση μιας συγχρηματοδότησης και σε χώρες όπως η Ελλάδα έχουμε και μια συμφωνία που για πρώτη φορά φέτος θα τεθεί σε εφαρμογή για διεθνή ενίσχυση υπό τη μορφή πιστώσεων και που μέρη των πιστώσεων αυτών πάνε και στην συγχρηματοδότηση έργων των διαρθρωτικών ταμείων που σημαίνει ότι για φέτος για πρώτη φορά θα εξαντλήσουμε τον σχεδιασμένο προϋπολογισμό με κοινή βοήθεια και αυτό θα συνεχιστεί και του χρόνου. Στον δημόσιο τομέα λοιπόν αρχίζει πάλι να υπάρχει κάποια κίνηση. Η δυσκολία βέβαια είναι ακόμα στον ιδιωτικό τομέα. Α, τώρα, μεταβατικές περιφέρειες. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες ξεφεύγουν πλέον από την ζώνη του 75% που για άλλους λόγους ήταν κάτω από το 75% Υπάρχουν στην Ευρώπη 16 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε περιφέρειες της ζώνης μεταξύ 75% και 90% σε τρόπο ώστε να φαίνεται να χρειαζόμαστε μια ενδιάμεση κατηγορία για να διασφαλίσουμε τα επιτεύγματα αυτά αλλά ταυτόχρονα να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την βελτίωση του επίπεδου ευημερίας. Ο στόχος, όπως είπα και πριν, είναι η τελική σύγκληση. Σύμφωνα και με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων, οι πληρωμές να γίνουν τρόπο περίπου ισότιμος τα 7 χρόνια με μια καμπύλη η οποία σιγά σιγά να μειώνεται, να φθήνει, να είναι ένα είδο ομαλής προσγείωση. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πέντε λεπτά μονάχα τώρα για την στατική του Δούναβη. Ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Δεν το συνηθίζετε αλλά το ότι δεν, μας δώσατε το λόγο το θεωρώ ότι είναι διάκριση σε βάρος της GUNGL και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χύπνερ, μακάρι να είχα περισσότερες δυνατότητες στα χέρια μου και να μπορούσα την ημέρα των 24 ωρών να την κάνω 48. Αλλά σας υπόσχομαι, εάν ο ε, κύριος Επιτρόπος τελειώσει νωρίτερα, θα σας δώσω πάλι τον λόγο. Εκτός αν θέλετε καλύτερα να είστε πρώτος στη λίστα του Ιανουαρίου. Αλλά δυστυχώς δεν έχω περισσότερε δυνατότητε. Yeah, ο επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ θα ξαναέρθω τον Γενάρη και θα προσπαθήσω να δίνω και συντομότερες απαντήσεις. Στατηρική του χώρου του Δουνάβεως. Χθες στην Κομισιόν εγκρίναμε το σχέδιο της στρατηγικής μαζί και με σχέδιο δράσεως με στόχο ώστε τον Απρίλη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων υπό Ουγγρική Προεδρία να εγκριθεί η στρατηγική αυτή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλέον του Ιουνίου από τους αρχικούς κατών κυβερνήσεων ώστε στον χώρο του Δούναβη που είναι και ο πιο ο, ο ποταμός ανά τον κόσμο που έχει την περισσότερη κίνηση και με 10 χώρες που ε, βρέχονται από αυτόν από τις οποίες περνάει μέσα. Και με τις τρεις μεγάλες θρησκείες, με σημαντικές βέβαια οικονομικές ανισότητες, αλλά και με εκ του λόγου τούτου τεράστιο δυναμικό, θα υπάρξουν τέσσερα μεγάλα κεφάλαια και ένδεκα προτεραιότητες. Τα κεφάλαια είναι αφενός το θέμα της πλοημότητας του Δούναβη, που σε σχέση με τον Δούναβη έχουμε ένα δυναμικό το οποίο ε, ε, το εκμεταλλεύονται μέχρι 3 έως 6% σε σχέση με τον Ρήνο, επαναλαμβάνω. Βελτίωση και της ε, περιβαλλοντικής κατάστασης και της ποιότητας των νερών αλλά και της βιοπικιλότητας στον χώρο του Δούναβη. Έχουμε τώρα και ένα δεύτερο πυλώνα που έχει σχέση με την ανάπτυξη ε, των ανθρώπινων πόρων, του λεγόμενου capacity building και όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος όπως για όλες τις μακροοικονομικές στρατηγικές ισχύει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ούτε επιπρόσθετοι κανόνες, ούτε επιπρόσθετη γραφειοκρατία, αλλά ούτε και επιπρόσθετα κονδύλια, διότι θεωρούμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι τα εφιστάμενα κονδύλια από τα διαθωτικά ταμεία μαζί με τα χρήματα των προενταξιακών πιστώσεων κτλ. να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδοθεί προστιθέμενη αξία που σημαίνει να βασιστούμε αποκλειστικά να ρίξουμε το ιδιαίτερη προσπάθεια ειδικά σε έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν με συνεργασία πλειώνων περιφερειών για παράδειγμα στην βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, στην πλοημότητα, στην οικονομική ανάπτυξη, στην ε, συνεργασία σε τα πολιτιστικά. Αυτά όλα γίνονται μόνο με συνεργασία. Το 2012 θα υποβάλουμε την πρώτη ενδιάμεση έκθεση και αυτά είναι εν ολίγης τα στοιχεία τώρα της στρατηγικής του χώρου του Δουναβή. Η ιδέα αυτή έχει προκαλέσει και στις χώρες μέλη σημαντική ευφορία. Μέχρι τώρα έχουν ε, δημοσιευτεί 800 γνωμοδοτήσεις στην ε, πορεία των μέχρι τώρα διαβουλεύσεων και αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα. Δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια στην Ευρώπη που να μην επιθυμεί να συμμετέχει σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα στο Δούναβι και ίσως μετά μπορεί να καταστεί εφικτό ένα επόμενο βήμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Ελπίζω να συμφωνήσετε για το Δούναβι. Το θέμα του Δούναβι τον Ιανουάριο νομίζω ότι ο κύριος Αγκουράκης θα μπορούσε να υποβάλει την ερώτηση τώρα αλλά έχει αποχωρήσει. Θα είναι ο πρώτος ομιλητής τον Ιανουάριο Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, στην ατζέντα μας γενικά ε, από τώρα μέχρι το καλοκαίρι. Εάν βρούμε επιπρόσθετο χρόνο θα προβάλλουμε, θα οργανώσουμε δύο συναντήσεις το επόμενο έτος. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα ε, θα δούμε το θέμα ΚΡΕΛ. Το θέμα 5 στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα υπαριθμών 5. Κάναμε αλλαγή μεταξύ του 4 και 5. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα η Κωνσταντσε Κρέλ να μας μιλήσει για την έκθεσή της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη σχετικά, διότι εκτός των όσων είχα αναπτύξει στην πρώτη συζήτηση δεν έχω βέβαια να προσθέσω σε αυτά πάρα πολλά πράγματα πριν να στείλω το έγγραφό μου στην μετάφραση είχα συζητήσει και με τους σκιώδεις εισηγητάς και εισηγητρίας ώστε στο μέτρο του δυνατού να περιλάβω και ιδέες των ε, προσώπων αυτών. το σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Αυτό καθίσταται σαφέ σε ορισμένες παραγράφους για το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης. Νομίζω ότι για την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και για τον κύριο Γκαρίγα, τον εισηγητή, είναι σημαντικό να καταστήσουμε και πάλι σαφή την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Μαζί με τους κοιόδης συγητάς διεξαγάγαμε συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να περιληφθούν άλλες προτεραιότητες. Ωστόσο νομίζω ότι είναι σημαντικό η γνωμοδότησή μας να περιοριστεί στις πιο σημαντικές προτεραιότητες. Και νομίζω αυτές που έχουμε περιλάβει παλαιότερα σε ψηφίσματά μας. Σημαντική επίσης είναι η επισήμανση στη γνωμοδότηση ότι θέλουμε το Περιφερειακό Ταμείο να, παραμείνει μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής όπως έδειξε άλλωστε ε, και η ίδια η συζήτηση που μόλις διεξαγάγαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό στο παρελθόν είχαμε ολοκληρώσει επιτυχώς τη συζήτηση για τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική πολιτική που θέλουμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό το περιλαμβάνω και στην γνωμοδότησή μου, διότι πράγματι διακόπτει η κυρία Κρέλη γιατί γίνεται θόρυβος. Σας παρακαλώ λοιπόν. Διότι πρόκειται για θέμα το οποίο είναι σημαντικό για την εδαφική συνοχή και συχνά θεωρείται ως παράρτημα περισσότερο. Γι' αυτό το περιλαμβάνω τώρα ευθέω στη γνωμοδότησή μου. Πρέπει να φροντίσουμε βέβαια να καταστεί σαφές ότι θέλουμε η πολιτική συνοχή να είναι στη διάθεση όλων των περιφερειών, να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις, δεν ξέρω ποιου χαρακτήρα. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν ακόμα και αυτή δεν έχει καταλήξει και ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμα διαπραγματεύσεις Εγώ συντάσω και την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Σούρε, επομένως είναι κάποια στιγμή θέμα χρημάτων, κονδυλίων. Να δούμε λοιπόν ποια πράγματα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και να δηλώσουμε καθαρά ότι θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να υλοποιηθεί μοναχά με επίπεδο κονδυλίων που θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο επίπεδο που διαθέτουμε σήμερα και δεν πρέπει να μειωθεί. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να δηλωθούν από πλευρά τη Επιτροπή μα με ξεκάθαρο τρόπο και έτσι τα έχω γράψει κιόλας μέσα. Σε ό,τι αφορά την διάρκεια της μεσοπρόθεσμης του μεσοπρόθεσμου μάλλον δημοσιονομικού σχεδιασμού γράφω ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ετών εάν κάποια στιγμή καταλήξουμε να είναι 10 χρόνια ή δύο φορές από 5 χρόνια θα είναι και αυτό ίσως ένα αποδεκτό αποτέλεσμα αλλά πάντως θέλω να περιλάβουμε την μνήμα ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ετών. Ο κ. Γκαρίγα, ο οποίος στο τελευταίο του έγγραφο, στη τελευταία του ε, σχέδιο της εκθέσεως δεν έχει καν περιλάβει την δυνατότητα ότι θα μπορούσε να είναι 7 ετών, ελπίζω να δεχθεί ότι για την πολιτική συνοχή τουλάχιστον θέλουμε τουλάχιστον 7 χρόνια. Αυτό που δεν είναι σαφές για μένα είναι πού θα καταλήξει η συζήτηση εφόσον υπάρξουν εξαιρέσεις για την πολιτική συνοχή, για την πολιτική έρευνα και ούτω καθεξής, που είναι συνολικά αυτές οι ξεχωριστές πολιτικές περίπου τα 2 τρίτα του προπολογισμού. Πώς θα είναι δυνατόν για αυτές τις πολιτικές να προπλευθούν διάρκειες των δύο, φορά, δύο φορές πέντε ετών, ενώ για τον υπόλοιπο προπολογισμό που θα καταληξει η συζητηση εφοσον υπαρξουν εξαιρέσει για την πολιτικη συνοχη για την πολιτικη ερευνα και ουτω καθεξης που ειναι συνολικα αυτες οι ξεχωριστες πολιτικες περιπου τα δυο τριτα του προπολογισμου πως θα ειναι δυνατον για αυτες τις πολιτικες να προπλευθουν διαρκειες των δυο φορα φορες πεντε ετων ενω για τον υπολοιπο προπολογισμο που θα ειναι το ένα τρίτο μόνο, πέντε ετών. Αυτό δεν το ξέρω. Θα δούμε ε, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και στην Επιτροπή ΣΟΥΡ. Κάτι που περιέλαβα επίσης στην γνωμοδότησή μου είναι ότι εμείς είμαστε ο μοναδικός τομέας πολιτικής και στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 περιλαμβάνουμε όλα τα τμήματα της πολιτικής αυτής, τη βιωσιμότητα, ε, την ευφύ ανάπτυξη και ούτω καθεξής, ότι είμαστε και κατά της τομεοποίησης της πολιτικής συνοχής, ότι καθιστούμε σαφές ότι στους τομείς αυτούς μεταφορές, συγκοινωνία, τομέας έρευνας, βλέπουμε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει επιτυχίες στη δημιουργία απασχόλησης και ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν μαχά μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής συνοχής και όχι εφόσον αυτή σπάσει σε τομείς Επίσης ε, επισημαίνω και πάλι στη γνωμοδότησή μου ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται εκ του αποτελέσματος, ότι χρειάζονται απλοποιημένες διαδικασίες ή δυνατόν ενιαίες διαδικασίες που να ισχύουν και για άλλους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε μια πιο αποδοτική χρήση των κονδυλίων, το καθιστώ και αυτό σαφές, και ελπίζω οι προτάσεις αυτές που κάνω να απηχούν τα βασικότερα θέματα που είχε συζητήσει η <clears throat> Περιφερειακή Επιτροπή και στις συζητήσεις της. Και αναμένω τώρα με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις των συναδέλφων μου. Τόμας Ντόιτς, σκιώδης συγητής του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη ε, δυνατότητα να λάβω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, ως σκιώδης από το ΕΛΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κωνσταντσε Κρέλ για την ενδιαφέρουσα εισήγησή της και αυτή την ε, ε, πρόταση που είναι μια ενδιαφέρουσα και ποιοτική πρόταση. Επίσης θα ήθελα να την ευχαριστήσω διότι είναι διατεθειμένη να, ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί με όλους τους σκιώδεις. Ήταν υποδειγματική η συνεργασία και οι περισσότερες τροπολογίες έχουν ενταχθεί στο κείμενο που έχετε ενώπιόν σας. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι ότι ως προς τα περισσότερα στοιχεία βασίζεται στην συνένεση αυτή η πρόταση, άρα μπορούμε εύκολα να την υποστηρίξουμε. Παρόλα αυτά, θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ορισμένα σχόλια και να τονίσω ορισμένα θέματα τα οποία έθιξε ήδη η εισηγήτρια προηγουμένως ή τώρα στην παρουσίασή της σήμερα το πρωί. Καταρχήν νομίζω ότι στο σημείο 15 της έκθεσης θα πρέπει να αποσαφινιστεί κάπως η διατύπωση και να πούμε ότι οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για, στο στον τομέα των ταμείων ε, συνοχής, ιδιαίτερα ως προς τα κονδύλια που δεν έχουν δαπανηθεί. Θα πρέπει δηλαδή να διασαφηνίσουμε κάπως την ε, παράγραφο 15, να αλλάξουμε τη σύνταξη της πρότασης και θα υποβάλουμε μια τροπολογία για το θέμα αυτό. Σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν από τον Επίτροπο την προηγούμενη μια μισή ώρα περίπου, θα ήθελα να πω ότι η στρατηγική 2020 είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτική σύνοχης που είναι μία από τις πλέον επιτυχείς πολιτικές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τολμώ να πω ότι υπάρχει συνένεση και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο ότι δεν μπορούμε να εξισώσουμε τη στρατηγική 2020 και την ε, πολιτική συνοχής. Γιατί η στρατηγική 2020 αφορά κάτι παραπάνω από μια πολιτική συνοχής. Και η πολιτική συνοχής δεν θέλει μόνο να προσδώσει νόημα στην ε, στρατηγική 2020. Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στην ΜΕΝ και τη ΔΕ. Θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση ότι η περιφερειακή πολιτική κάθε αυτή δεν ε, θα πληρώσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Συμφωνώ με τη βελτίωση του ανταγωνισμού. Υποστηρίζω την πρόταση της συναδέλφου. Θα ήθελα όμως να καταστήσω σαφές στο κείμενο ότι στην περίπτωση των περιφερειών βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Θα πρέπει να ισχύσουν διαφορετικά μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες των μεμονωμένων περιφερειών. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε μια συσταλτική ερμηνεία κάτι το οποίο δεν έκανε ούτε η συγγήτρια. Τώρα ο σύνδεσμος αυτός μεταξύ κοινωνικού ταμείου και πολιτικής συνοχής, αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη την ε, τροπολογία μου που μιλά για λειτουργική ολοκλήρωση, δηλαδή έμπρακτη συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έτπα καθώς και πολιτικής συνοχής. Τέλος, δύο ερωτήσεις. Πρόκειται για ερωτήματα που θίγησαν και την προηγούμενη φορά. Το ένα αφορά την αιρεσιμότητα, που είναι ένα κρίσιμο θέμα. Συμφωνώ με την προσέγγιση με τη Ρουμάνα συνάδελφο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αιρεσιμότητα ως μορφή κύρωσης. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό με τον Επίτροπο τον Ιανουάριο για να δούμε πώς θα ισχύσει η αρχή της αιρεσιμότητας και κατά πόσο ισχύει μόνο για την πολιτική συνοχής ή, και, εφαρμόζεται και σε άλλες πολιτικές. Τέλος, θα ήθελα να αποβάλω και ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο αναφέρουμε σε κάθε έκθεση, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι ότου τεθεί σε εφαρμογή. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές τα τρία θεσμικά όργανα ε, πολλές φορές μοιάζουν με ένα παιχνίδι παιδιών. Δηλαδή μου θυμίζει το χαλασμένο τηλέφωνο γιατί μέχρι ότου φτάσει το μήνυμα στο τέλος της γραμμής είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Δηλαδή χάνεται το μήνυμα μέσω μεσαζόντων. Αυτή την εντύπωση έχω γιατί μιλάμε για την ανάγκη απλούστευσης και αυξάνουμε κατ' ουσίαν τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το πλαίσιο, λιγότερη γραφειοκρατία, και λιγότερο δαπανηρή εφαρμογή. Και χαίρομαι για την έκθεση. Ο Φρανσουά Αλφονς είναι ο επόμενο ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ Κωνσταντζα και για τη δουλειά σου και για τη συνεργασία σου για τα βασικά σημεία. Πολλά από αυτή την έκθεση μας αρέσουν, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς τις πολιτικές συνοχής διευκρινίζοντας διότι αυτό θα ήταν τελικά ε, μέχρι και αντίθετο με τη συνθήκη της Λισαβόνας, διότι η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει για τη χωροταξική συνοχή και να αμφισβητούμε εμεί σήμερα στην περιφερειακή της διάσταση θα ήταν σαν να αντιβαίναμε τη συνθήκη. Επίσης, θα πρέπει να προσαρμοστούμε όχι μόνο στις νέες προκλήσεις αλλά και στις νέες πραγματικότητες. Μας το είπε και ο Επίτροπος. Ο στόχος ένα σήμερα αφορά 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους έναντι των 170 της προηγούμενης περίοδου. Και θέλουμε ταυτόχρονα να διατηρήσουμε και το δημοσιονομικό επίπεδο. Η φυσική απόφαση, η λογική απόφαση που θα μπορούσε να λάβει ένας νομοθέτης ήταν εφόσον καλύπτονται λιγότερα εκατομμύρια τότε μειώνουμε τον προπολογισμό. Αυτό όμως στρεβλώνει την πραγματικότητα διότι πέρα από την... Ε, ε, πέρα από αυτήν την αλλαγή υπάρχει και οικονομική κρίση η οποία τελικά ε, αποδυνάμωσε πολλές ε, περιφέρειες θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε εμείς με τον ίδιο προϋπολογισμό ούτως ώστε να μην τις λυγίσουμε ακόμη παραπάνω. Θα έπρεπε λοιπόν να ορίσουμε, όπως είπε ο Επίτροπος, έναν ενδιάμεσο στόχο να πούμε ότι η σκοπιμότητα μιας πολιτικής συνοχής δεν είναι να σταματήσει στο 75%. Πρέπει να προχωρήσει πιο πέρα. Γιατί 75% για τους στοχότερους τι σημαίνει 200% για τους πιο πλούσιους. Η ψαλίδα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στη χωροταξική συνοχή όπως μας το απαιτεί η συνθήκη της Λισαβόνας. και προγραμματίζουμε την πολιτική μας μακροπρόθεσμα και βγαίνουμε από αυτή τη λογιστική παγίδα που λέει ότι εντάξει λιγότεροι πολίτες εποφελούνται άρα μικρότερος προπολογισμό. Όχι. Πρέπει να κρατήσουμε τις πιστώσεις διότι ο στόχος μας είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Αυτά λοιπόν. Τώρα για ένα άλλο θέμα ουσίας είναι να συνεισφέρουμε με περισσότερες πιστώσεις και μεγαλύτερη υποστήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία. Αναφέρεται αυτό και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να καταστεί ένας στόχος ε, πιο ορατός ε, για τις πολιτικές ε, συνοχής. Διότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα πρέπει να έχει αυτήν την ε, να δίνει αυτή την εικόνα στα μάτια των πολιτών, να την αναγνωρίζουν σε ευρωπαϊκή πολιτική, να αρχίσει να κινείται αυτή η πολιτική, να υλοποιεί πράγματα και να την αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτά για τα ουσιαστικά και συμφωνώ με την Κωνσταντζα για τη διάρκεια, για το χρόνο. Εμείς ε, μπαίνουμε σε μία λογική που πρέπει να αλλάξει που θα πρέπει πέρα βέβαια από τα πέρα από τις ε, διάφορες βιαστικές αποφάσεις ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε, μια μεγαλύτερη, σε, ένα μεγαλύτερη, σε ένα μεγαλύτερο προγραμματισμό. Δεν μπορούμε όμως από την άλλη μεριά και με αυτό το 5 συν 5 να ε, περιμένουμε για την ε, συνοχή τόσο πολύ 5-5 δηλαδή μας κάνει 10, περνάμε από τα 7 στα 10. πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα αντίδρασης για να προσαρμοζόμαστε στις νέες ε, πραγματικότητες. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με την ε, Κωνσταντζα για αυτά τα τελευταία, 7 χρόνια. Και το να έχουμε κυρώσεις για κυβερνητικές πολιτικές εμείς συμφωνούμε γύρω από προγράμματα ξέρουμε ότι είναι χρήσιμο για την Ευρώπη, χρήσιμο για την περιφέρεια ένα πρόγραμμα και του αφαιρούμε τελικά τις πιστώσεις όταν ξέρουμε ότι λειτουργεί πολύ καλά. Λοιπόν, δεν είναι λογικά όλα αυτά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να δούμε πώς θα συμφωνήσουμε για όλες αυτές τις προτάσεις. Ο Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Εγώ νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν για το 90%. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το σημείο 5 και πιο συγκεκριμένα για τη στρατηγική διότι καλύπτονται τα πάντα και οι πολιτικές που θέλουμε να ενθαρρύνουμε και όλα. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Τώρα για την ε, ε, κάλυψη την, στον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του θα πρέπει να είμαστε πιο αυτοκριτικοί ως περιφερειακή πολιτική. <coughs> Εμείς Μήπω το 5 συν 5 δεν θα ήταν καλύτερα για μα για να είμαστε πιο αξιόπιστοι διότι αυτό το 7 μου φαίνεται μένα λίγο σύντομο. Δεν θα ήταν ίσως μια ευκαιρία για μας. Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτούμε, θα το άφηνα εγώ ανοιχτό όλο αυτό και θα κοίταγα να ζητήσω τις σχετικές συμβουλές να, να, μας συμβουλέψουν, να μας πούνε γιατί δεν μπορούμε εμείς τελεσίδικα να πούμε 7 χρόνια, πρέπει να εμβαθύνουμε. Δεν καταλαβαίνω εγώ ορισμένου συναδέλφους που λένε ότι δεν πρέπει να, να, να πειράζουμε τα ταμεία συνοχής όταν φύγονται οι αρχές ε, της σταθερότητας. Μα ξέρουμε πολύ καλά όμως ποιες είναι οι χώρες. Είναι πάντα ίδιες. Και η Κομισιόν μας το λέει πάντα. Μπορούμε εμείς να πούμε με πλήρη συνείδηση ότι οι χώρες οι οποίες συνειδητά δεν τα κριτήρια του Συμφώνου σταθερότητα, μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούν σωστά τα, ε, τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Εμένα η απάντησή μου είναι όχι. Γίνεται κακή χρήση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε αυτό το ειδικό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε συνείδηση αυτών των δυσκολιών και να κοιτάξουμε να βρούμε μία απάντηση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Κρέλ κατά ένα 98%. Χαίρομαι διότι στην γνωμοδότησή της ασχολήθηκε με την πολιτική συνοχής κατά ένα πολύ σωστό και συνετό τρόπο. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές, να είμαστε απόλυτα σαφείς. Μέχρι τώρα στην ε, Επιτροπή. Οι συζητήσεις μας ήταν πολύ θεωρητικές, αλλά νομίζω ότι ήρθε πια η ώρα για να ε, μετατρέψουμε τη θεωρία σε πράξη και νομίζω ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τον ε, Ιανουάριο θα πρέπει να μιλήσουμε για το προκείμενο και γι αυτό, θα, γι' αυτό είναι και η κατάλληλη στιγμή για αυτή τη γνωμοδότηση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εκείνοι που θα πρέπει να εργαστούν με τα, μία συνοχή, με τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να λάβουν υπόψη την επταετία που είναι μια, ε, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε με τις χρονικές περιόδους, αλλά θα πρέπει να επιμερίσουμε το χρόνο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Στην, ως προς την πολιτική συνοχής γενικότερα υπάρχει τάση στις συζητήσεις μας να επανεθνικοποιήσουμε ορισμένους τομείς και να δώσουμε τομεακή διάσταση σε άλλα θέματα. Είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κοινοτική πολιτική, όχι λιγότερη. Και ο πλέον λογικός τρόπος να το επιτύχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά την ίδια την πολιτική συνοχής. Πολλοί μιλάνε για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Αυτή τη συζήτηση την προθήσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητήσαμε το θέμα και με την Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι οι συζητήσεις δεν έφτασαν μέχρι το ευρύ κοινό. Ο συνάδελφος είπε ότι οι ιδέες γίνονται πραγματικότητα όταν ε, φτάσουν στις μάζες και η στρατηγική 2020 θα πρέπει να ενταχθεί στις περιφέρειες, θα πρέπει πρώτα να φτάσει στις περιφέρειες. Αυτό το συζητήσαμε και με τον Επίτροπο και επ' αυτού πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ε, μία άρση αυτής της τροχοπέδης που είναι τα, τα κράτη Πολλές φορές γίνεται ανεπαρκής χρήση ε, πόρων ή δεν γίνεται σωστή χρήση από τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να επιτελέσουμε μεγάλο όγκο εργασίας για να επιτύχουμε μια καλύτερη εφαρμογή. Και βεβαίως ο καθένας στη χώρα του θα πρέπει να ορίσει τα του οίκου του. Πρωτίστως, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ε, εισαγάγουμε πολλά στοιχεία, θα πρέπει να αρκεστούμε στις προτεραιότητες και μετά τα άλλα μέλη της Επιτροπής θα μιλήσουν υπέρ της ε, πολιτικής συνοχής. Ε, thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι προς τον συνάδελφο που αποχώρησε γιατί είπε ότι δεν είχε το λόγο και γίνεται ε, διάκριση ε, κατά μερικών. Έχει δικαίωμα να έχει όποια γνώμη θέλει, αλλά όταν υπάρχουν ε, πέντε λεπτά και 11 ομιλητές θα πρέπει να αποφασίσει η πρόεδρος, δεν πρέπει να κατηγορείται. Σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια, αυτό το 5 συν δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μπορούμε να έχουμε 7 συν 3, αν θέλετε μία ε, διετή εντολή ή δύο εντολές. Αυτό συζητιέται εδώ και πολύ χρόνο. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουμε. Εγώ προτιμώ ε, ένα επταετές πλαίσιο και όχι πενταετές. Ο Τόμας επίσης αναφέρθηκε στο θέμα της απλούστευσης. Δηλαδή καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες και χάσαμε πολύ χρόνο ε, μέσα στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών χωρίς να τα θέσουμε όλα αυτά στην ε, πράξη. Θα πρέπει να δούμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί, να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, νέες υποδομές. Άρα ε, απλούστευση βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε με μία αδαπανηρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιμερίσουμε αυτή την ε, πολιτική μας στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Κρέλ κατά ένα 95-96%. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των διαφόρων σχεδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χρηματοδότηση από διαφορετικά ταμεία. Να δούμε δηλαδή πώς ε, ε, είναι αλληλένδετα αυτά τα σχέδια. Όπως είπε και ο κύριος Κέλλη, θα πρέπει να επιμείνουμε ως προς το εξής. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα πρωτίστως για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται επαρκής χρήση των μέσων. Επίσης έχει μεγάλη σημασία η ευελιξία γιατί σε μία τέτοια δημοσιονομική περίοδο ίσως μπορούν να υπάρξουν πολλές αλλαγές. Επίσης θεωρώ ότι εάν λάβουμε υπόψη την παρούσα κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε το επίκεντρο προσοχής μας, δηλαδή να δούμε την οικονομική διάσταση ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών και να δούμε πώς θα αναπτυχθεί και αυτή η οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών. Όμως ε, δεν υπάρχει αυτή η δημοτική πτυχή όπως θα θέλαμε, δηλαδή η συμμετοχή των τοπικών αρχών. Αυτά συζητούνται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και θα πρέπει αυτό να αναφερθεί και από την έκθεση κάθε. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι θα πρέπει να δούμε ποια διάσταση δίνεται σε αυτήν την εργασία και πώς διαδίδεται αυτή η εργασία. Και εδώ μιλώ για την έμπρακτη πορεία μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα μέτρα, όχι για δημοσιοποίηση απλώς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα διοχετευτούν τα κονδύλια αυτά και ε, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Κρέλ. συμφωνούμε κατά 90% με τις εκτιμήσεις της. Χαίρομαι και για ορισμένε ιδέες που ακούστηκαν. Επιθυμώ επίσης να τονίσω ορισμένα πράγματα. Ιδίως την ε, εδαφική διάσταση που ελπίζω να μην αποκαλύψει νέες αδυναμίες η πολιτική συνοχής είναι από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την συνέχιση της επιτυχίας αυτής και δυνατόν και την μεγεθυνσή της. Όταν μιλήσαμε για επικουρικότητα, ε, για τον ρόλο όλων των συμμετεχόντων επιπέδων κρατών, περιφερειών κλπ. Είναι σωστά αυτά. Εγώ θέλω να θυμίσω ωστόσο και την ισορροπία ανάμεσα στην μεγάλη πόλη, την Κομόπολη και, το, ε, και την Ήπεθρο. Βέβαια, η μεγάλη πόλη θα παίξει σημαντικό ρόλο γιατί είναι ο σημαντικός πόλος, ο κινητήρας της ε, ανάπτυξης. Όταν μιλούμε όμως για τα υπόλοιπα 155 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίων που ζουν σε άλλες περιφέρειες ή ε, στην Ήπεθρο δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε αυτά διότι θα οδηγηθούν σε μειονεξία. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, πρέπει να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις ώστε αυτή, αν με επιτρέπετε, η μακροισορροπία να μην ανατραπεί ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις, τις κομοπόλεις και την Ήπεθρο. Ε, τώρα έρχομαι στον κύριο Ντόιτς που είπε σωστά ότι εδώ μιλούμε και για κυρώσεις, για τιμωρητικούς μηχανισμούς και για νέους κανόνες. Αλλά πρέπει να μην λησμονήσουμε ότι χρειάζεται και μια απλοποίηση όλης της διαδικασίας στην πολιτική συνοχή. Πάλι που αναφέρεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι για να μην χάσουμε την ισορροπία, τη συνολική ισορροπία, όπως είπα και πριν. Εν τέλει, και συμφωνώ πάλι με την πρόταση Deutsch, δηλαδή για τις δαπάνες που μπορούν ακόμη να κατανεμηθούν στις διάφορες χώρες μέλη και που νομίζω ότι για κάποιο διάστημα μπορούμε να διατηρήσουμε τον κανόνα νη συν 2 και νη συν 3 εφόσον δεν ε, ε, υπάρξουν άλλες διευρύνσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη συνεργασία με τη συνάδελφο Κωνσταντς και θα ήθελα να ολοκληρώνω λέγοντας θα θέλαμε να δούμε αν θέλουμε μάλλον να δούμε επιτυχία θα πρέπει να εγκρίνουμε τις παραγράφους 1 19 της εκθέσεως είναι ίσως ε, δυνατόν να βελτιώσουμε κάποιες παραγράφους αλλά καμία δεν μπορούμε να διαγράψουμε. Η παράγραφος 10 για μένα είναι σημαντική. Μια ε, επιτυχημένη ε, πολιτική συνοχής χρειάζεται χρηματοδοτικά μέσα. Ενώ πάνε τώρα να τα μειώσουν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Είπε ο Επιτροπός ότι αν περικοπεί ο προϋπολογισμός θα υπάρξουν αναλογικά επιπτώσεις για, σε βάρος όλων των χωρών αλλά υπάρχει διαφορά. Εάν τα χρήματα αφαιρεθούν από περιφέρειες όπου το ελάχιστο εισόδημα είναι 1.600 ευρώ το μήνα ή από την ε, περιφέρεια ή την Ήπεθρο όπου υπάρχουν χώρες και περιφέρειες όπου το μέσο εισόδημα είναι της τάξης των 120 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν τέτοιες χώρες και τις περιφέρειες στην Ευρώπη η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται στο Συμβούλιο. Ο προπολογισμό έγινε το εργαλείο για την άσκηση πολιτικής, μικροπολιτικής. Για τον λόγο αυτό πρέπει να πιέσουμε τις χώρες μέλη να αντιληφθούν ότι εάν δεν προβλεφθούν αρκετά κονδύλια θα πληγούν οι φτωχότερες χώρες πρωτίστως. Σε ό,τι αφορά την περίοδο σχεδιασμού και σε σχέση με την στατική 2020, προσωπικά πιστεύω ότι τα 7 χρόνια είναι η καλύτερη επιλογή. Sophie, I'm using your name not properly. I'm saying Sylvie all the time, but I think Sophie. Oui. Σε λέω Σίλβιο, αλλά σε λέει Σοφία. Ναι, ναι, ακριβώς. Και ε, Σοφία, θα πει Σοφία και θέλω να το κρατήσω το όνομά μου. Ε, σχεδόν όλα υπόθηκαν για την ε, τόσο καλή δουλειά της κυρίας Κρέλ. Αλλά για το πρόγραμμα, για την περίοδο προγραμματισμού. Εγώ συμφωνώ με τον Μάριους Πίπερ και την θέση του Αλφόνση. Εφτά χρόνια μου φαίνεται μια κατάλληλη, είναι μια σωστή περίοδος για μένα. διότι υπάρχει και μία συνοχή των δράσεων μετα μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Αλλά αυτό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο σωστός χρόνος πριν. Δηλαδή, εμείς έχουμε ας πούμε το, το, το, το πρόγραμμα μέχρι το 2013, το οποίο το 2007-2013, το οποίο το επεξεργαστήκαμε το 2005, όπου η κατάσταση και η συγκυρία ήταν εντελώς διαφορετική, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τι θα γινόταν σήμερα. Θα έπρεπε λοιπόν, και το θεωρώ ενδιαφέρον, να προσαρμόζουμε τους κανονισμούς για την περιφερειακή πολιτική ανάλογα με τη συγκυρία, με την περίσταση η οποία αλλάζει 5 συν 5 ναι, αλλά υπό την επιφύλαξη ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ε, την ποιότητα της εργασίας της κυρίας Κρέλ. Μία απλή παρατήρηση. Είπα ότι η έκθεση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία να διευκρινίσουμε ορισμένες πολιτικές. μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την χωροταξική συνοχή, την αλληλεγγύη. Αλλά βάζει σε ανταγωνισμό τις περιφέρειες για την χρηματοδότησή τους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό και να ξεκαθαρίσουμε τι είναι χωροταξική συνοχή. Να μην υπάρχει αμφισημία ε, για ορισμένους όρους όπως είναι ο ανταγωνισμός, η συνοχή, η ελληνική. Αυτές είναι οι απλές παρατηρήσεις που ήθελα να διατυπώσω σχετικά με την έκθεση. Τελειώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Η Ελίζα το λόγο. Ε, και βεβαίω θέλω τον λόγο και μάλιστα η γραμματεία μου ένευσε καταφατικά ότι με είδε και με σημείωσε. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα. Διότι έχω συμμετάσχει και μία από τις συζητήσεις της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Έχω την εντύπωση για την ώρα ότι και οι δύο επιτροπές ζουν στον κόσμο τους. Και η μόνη δυνατότητα συνδιαλέξεως είναι οι πολιτικές ομάδες όπου συμμετέχουν τα διάφορα μέλη της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Είναι σαφές για μένα ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες έχουν διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά τη ε, διάρκεια της ε, προγραμματικής περίοδου. Και ε, κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ είπα εγώ καθαρά ότι δεν μπορώ να φανταστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πλειοψηφία του να ταχθεί τελικά υπέρ μόνο πέντε ετών για την πολιτική συνοχή. Όλοι οι βουλευτές έχουν και εκλογική περιφέρεια και βλέπουν στην πατρίδα τους πώς είναι τα πράγματα και τι θα σήμαινε αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια δημοκρατική βούληση από καιρού καθιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπέσουν οι δύο περίοδοι. Και μάλιστα σχεδόν σημειώθηκε πλειοψηφία στο προηγούμενο κοινοβούλιο υπέρ της ιδέας αυτής. Εγώ θεωρώ παράλογη την ιδέα να πούμε ότι δύο τρίτα του προϋπολογισμού να λειτουργήσουν σε 7 χρονη βάση και το 1 τρίτο σε 50 χρονη βάση. Και μάλιστα τα 2 τρίτα είναι μάλλον 3 τέταρτα στην πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Στην Επιτροπή Σούρε είπαν ναι βεβαίως υπάρχει επιτροπή Σούρε και όλες εδώ οι επιτροπές εκπροσωπούνται άρα δεν χρειάζεται να γίνουν παράλληλες ε, ε, συνεδριάσεις αλλά πραγματικά στην επιτροπή Σούρε τον τόνο υπαγορεύουν τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών σαν δίθεν να μην υπάρχουν οι άλλοι. Ε, γι' αυτό και παρακαλώ την Πρόεδρο να ξανασκεφτεί πώς είναι δυνατόν να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί την ίδια ιστορία βλέπουμε και σε θέματα κατανομής της ε, πολιτική συνοχή. Μάλιστα εδώ έχουμε και απόφαση του Κοινοβουλίου, δηλαδή το ψήφισμά μας του Νοεμβρίου ή τελών, τελών Οκτωβρίου, που λέει καθαρά ότι θα πρέπει να παραμείνει ως ανεξάρτητη πολιτική η πολιτική συνοχής και μόνον τότε θα είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει η πολιτικη συνοχη και μονο τοτε θα ειναι σιγουρο οτι θα μπορεσει να λειτουργησει η ευρωπη του 2020. Όμως στην Επιτροπή Σούρε μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να σπάσει σε τέσσερα κομμάτια. Εγώ το θεωρώ παράλογο αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται η συζήτηση αυτή όμω. παράλληλα. Πρέπει και σύντομα να υπάρξει μια διευκρίνηση. Διότι προ τα έξω δίνουμε απολύτως συγκεχημένη εικόνα. Και δεν θα μπορούμε να εμφανιστούμε στις περιφέρειες αν ακούσουν οι άνθρωποι τι συζητούμε εκεί και κυρίως ότι δεν προχωρούμε ενώ ο χρόνο περνά. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα, Κωνσταντσε, αυτά τα σημεία διαφωνίας να τεθούν στις διαπραγματεύσεις ώστε να καταστούν ξεκάθαρες οι ε, διαφορές. Να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι διατυπώσεις, πιο αυστηρές οι διατυπώσεις. Να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή των πέντε ετών στην πραγματικότητα. Και ότι είναι σαφής η άποψη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. και να γίνει και μια συζήτηση έστω και μεταξύ δύο αντιπροσωπιών των δύο αυτών επιτροπών Περιφερειακής και Σούρε. Η ΔΕΜΗ, όπως είπα, η εργασία που κάνουμε κινείται παραλίλω και κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε αδίέξοδο. Κωνσταντζε. Ευχαριστώ για τις πολλές προτάσεις και ιδέες που έγιναν. Θα προσπαθήσω και η ίδια να υποβάλλω ορισμένε τροπολογίε. Δεν μου φάνηκε να υπάρχει καμία αμφιγνωμία. Σε ό,τι αφορά την διάρκεια, εγώ έχω γράψει 7 χρόνια που θεωρώ και λογικό και ότι έχει αποδείξει την αξία του, αλλά αφήνω ανοιχτή τη δυνατότητα να είναι και περισσότερο, δηλαδή δύο φορές πέντε χρόνια. μπορούμε να ξαναπούμε καθαρά ότι λιγότερο δεν είναι δυνατόν. Αλλά έχει δίκιο η κυρία Σουέντερ. Από τη δική μου πολιτική ομάδα γνωρίζω. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνει ας πούμε, μαχητική ψηφοφορία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ίσως είμαστε μισή-μισή. Αλλά η πρόταση να συζητηθεί από κοινού με την Σούρε είναι ενδιαφέρουσα. Διότι ακόμα και για λόγους δημοκρατίας έχω μάλλον ε, ε, με το, με το σύνθημα δημοκρατία δεν είμαι βεβαία ότι πρόκειται να γίνει τίποτα διότι δεν είμαι σίγουρη άλλωστε η αποχή από τις ευρωεκλογέ ήταν πολύ σημαντική σε όλες τις χώρες μέλη στην πραγματικότητα δεν ξέρω λοιπόν που θα καταλήγαμε αν κάναμε τέτοια προσπάθεια και μήπως στην πραγματικότητα μάλλον υποστεί πλήγμα η δημοκρατία στην Ευρώπη με μια τέτοια συζήτηση και γι' αυτό ότι είναι σωστό όπως βρισκόμαστε μέσα τώρα στην, στα μισά της, ε, της κοινοβουλευτικής θητείας όπου δεν υπάρχουν προεκλογικοί αγώνες, αλλά μπορεί κανεί πραγματικά να εγγύψει επί τη ουσία των θεμάτων. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν σωστό να ληφθεί η απόφαση αυτή. Βεβαίω είναι σε μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού τη ε, προγραμματική περίοδου και αυτό είναι σωστό να συζητηθεί. Αλλά μπορούμε, όπω είπε και η κυρία Σόιντερ, να κάνουμε μια συζήτηση με την κυρία Σούρε. Πάντω, εγώ την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλω το σχέδιο γνωμοδοτήσεως στον κύριο Γκαρίγα, εισηγητή της ΣΟΥΡΕ, διότι έχω μεγάλο ενδιαφέρον να περιλάβει στην δική του έκθεση έστω και τμήματα της γνωμοδοτήσεως Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι επιτυχής η προσπάθεια μου αυτή. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Όσον αφορά την τιμωρία, την επιφολή κυρώσεων, εγώ στην ουρομόδοτησή μου περιλαμβάνω μονάχα το θέμα εάν η πολιτική συνοχή μπορεί να θεωρηθεί ως κύρωση μόνο ε, στην περίπτωση που δεν τηρείται το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Για μένα είναι σαφές, εάν υπάρχουν, αν, υπά, καταχρήσεις των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κατάχρηση είναι κατάχρηση, η απάτη είναι απάτη. Αν θέλετε ωστόσο μπορώ να το περιλάβω για να... και για να φανεί καθαρά ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι μπορούμε σε κάποια σημεία να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες και ότι αυτές που έχουν περισσότερη ανάγκη πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο. Και να καταστήσουμε λέω και πάλι σαφές ότι για τις περιφέρειες οι οποίες εκπίπτουν των δύο κατηγοριών χρειάζεται μια ιδιαίτερη ρύθμιση. Δεν είμαι βεβαία διότι και με τις ερωταπαντήσεις σήμερα με τον κύριο Χάν δεν μου φαν, δεν είδα καθαρά εάν θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μια μεταβατική λύση, η ρύθμιση, εάν θα υπάρξει ένα νέο στόχος. Νομίζω πρέπει να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Ίσως βέβαια ήταν πρόημο ακόμα. Αλλά αναμένω με ενδιαφέρον ποιες ε, τροπολογίες θα υποβληθούν και θα δούμε. Αναμένω εν πάση περιπτώσει τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ ήδη για τη συνεργασία. Ευχαριστώ Κωνσταντσε. Το μόνο που θα πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών διότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Θα πρέπει να έχουμε χρόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα στις 16 Δεκεμβρίου γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Κωνσταντσε. Θα προτιμούσα λίγο συντομότερη προθεσμία, γιατί οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ήδη τι θέλουν και μέσα σε τρει μέρε μπορούν να γράψουν τα σχετικά κείμενα. Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα. Μετά όμω πρέπει να γίνει η εργασία, η, η περαιτέρω επεξεργασία. Και έχουμε και την μετάφραση που πρέπει να περιμένουμε να μπορέσω να υποβάλω και στα ουγγρικά το κείμενό μου στον κύριο ε, Ντόιτς. Θα προτιμούσα λοιπόν στις 14 6 το απόγευμα. Δηλαδή την Τρίτη. Λέτε γιατί την Τρίτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει η πρόταση από την Κωνσταντσε Κρέλ θέλει να έχει περισσότερο χρόνο να προσαρμόσει όλες τις τροπολογίες προτείνει τις 14 Δεκεμβρίου, δηλαδή την Τρίτη. στις 6 το απόγευμα, την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Τώρα προχωράμε στο σημείο 4. Ε, καλωσορίζω τους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να πω ότι στην ε, Επιτροπή Ρέτζιο την προηγούμενη φορά ζητήσαμε να μιλήσουμε για την ε, διασύνδεση μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και παροχής υπηρεσιών από ε, υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά μου δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη. Διαβάσατε τον τίτλο, μάλλον μπορείτε να τον αναγνώσετε κατά δύο τρόπους. Είτε καταφατικά, ότι υπάρχει δηλαδή διασύνδεση μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και υπηρεσιών γενικού συμφέρον, οικονομικού συμφέροντος, ή μπορείτε να το δείτε με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ε, αυτή η ε, διασύνδεση και προσπαθούμε να σας δώσουμε ε, ένα μία πρόορη ε, γνωμοδότηση σε σχέση με αυτές τις ε, μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, τη Λιέγη, καθώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Μιλάνο. Η συνεργασία έγινε μαζί και με το Βίλνιους, το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, Η Σίλβια ε, Βινιέτη και η Μπάρμπαρα Σάκ συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να πω ότι έχουμε πολύ καλή, είχαμε πολύ καλή σχέση με τους διαχειριστές της, ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ταμείων Συνοχής ε, ιδιαίτερα με την Έστερ Κράμερ. Υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία είναι να γίνει μία γενική συζήτηση για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μορφή παρουσίασης των ε, ε, υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και το οικονομικό είναι σε παρένθεση όπως βλέπετε. Θα πρέπει να σας πω προσωπικά ότι η οριοθέτηση του τι εμπεριέχεται σε μια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος ή υπηρεσία γενικού συμφέροντος, ε, αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν είναι και τόσο διαφανής ε, πάντα. Θα μιλήσω για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σαν ε, μια ευρύτερη, ως μια ευρύτερη κατηγορία και το περιεχόμενο αυτής της ενιολογικής βάσης των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και η σημασία για την περιφερειακή πολιτική είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Καταρχήν να δούμε την καθολική πρόσβαση ή προσβασιμότητα σε αυτές τις υπηρεσίες ε, από πλευράς χρηματοοικονομικής, οικονομικής και κοινωνικής και αυτό που έχει σημασία είναι και η ποιότητα των ε, υπηρεσιών καθώς και η προστασία των καταναλωτών ή τελικών χρηστών. Υπό μία έννοια λοιπόν Μιλάμε για διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές που εμπλέκονται. Και εδώ έχετε παραδείγματα από ε, μία μελέτη χαρτογράφησης από το CEP Δηλαδή, τι θεωρούμε ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Βλέπετε ότι μιλάμε για χρήσεις δικτύου, υπηρεσίες, ε, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητισμό, αναψυχή, κοινωνικοπολιτισμικές υπηρεσίες και άλλες. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαστάσεις, μία μακροδιάσταση διάσταση και μία μικροδιάσταση για να είμαστε σίγουροι ότι ότι συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά στην έκθεση, γιατί πρόκειται για μία ογκώδη έκθεση και δεν ξέρω αν θα τη διαβάσετε διεξοδικά, αλλά για να ρίξετε μια ματιά τουλάχιστον, θα ήθελα να αρχίσω με κάτι που δεν θα ξαναναφέρω. Σελίδα 113 βλέπετε έναν χάρτη με τουλάχιστον 27 σχέδια που την χάνουν υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ένα αναχώρα που μπορεί να σας δώσει μία γενική ιδέα για το πώς ε, δαπανώνται τα κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία στον τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Σε αυτό το δείγμα έχουμε περιλάβει και ορισμένα μικρά προγράμματα και άλλα μεγαλύτερης εμβέλειας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τα 27 προγράμματα, θα αναφερθώ σε ένα το οποίο σχετίζεται με το δεύτερο τμήμα του τίτλου, δηλαδή, δηλαδή διασυνοριακή συνεργασία. Κάθε φορά που το σκεφτόμαστε αυτό, αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία, θεωρούμε ότι πρόκειται για μία σιδηροτροχιά ή για έναν αγωγό φυσικού αερίου, κάτι τόσο ε, μεγαλειώδες. Δείτε όμως το σχέδιο στη σελίδα 147 που είναι το πρόγραμμα βαλτικών χωρών ε, στο τομέα της υγείας μέσω διαδικτύου, όπου στις, μεταξύ Σουηδίας, Λιθουανίας, Εστονίας, Νορβηγίας γίνεται μια ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τα εθνικά συστήματα υγείας. για τον τομέα της ε, ακτινολογίας και των υπερήχων. Δείτε στη σελίδα 152 της έκθεσης, όπου υπάρχουν δύο πιλωτικά σχέδια αυτού του προγράμματος, όπου διάφορα ε, νοσοκομεία μεταξύ Δανίας, Βίλνιους και Ταλίν ε, ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά πληροφορίες σε σχέση με ακτινολογικά δεδομένα έτσι ώστε να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα ε, της Δανίας όπου χρησιμοποιούνται οι γνώσεις παθολόγων από την Εσθονία και Λιθουανία. Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Για να κινηθούμε σε γενικότερα ζητήματα που περιλαμβάνονται, που εισάγονται εδώ, θα ήθελα να αρχίσω με κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό για σας, αλλά το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να τονιστεί. οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας, διότι βασιζόμαστε στο γεγονός ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση όπου και να βρίσκονται ό,τι εισόδημα και να έχουν δηλαδή ε, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Και ενώ γίνεται μία συζήτηση ευρωπαϊκής εμβέλειας σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο, μας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ολοκλήρωση της συζήτησης για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σε συσχετισμό με την περιφερειακή πολιτική. Αυτό μας ε, εκπλήσει διότι ε, πολλά από τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν να κάνουν με υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Άρα Όσοι εργάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο ασχολούνται με υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αλλά με μια διαφορετική προσέγγιση υπό μία έννοια. σε σχέση με εκείνους που εργάζονται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Άρα, οι δύο αυτές ε, τάσεις, ε, οι δύο αυτές συνιστώσεις τόσες, δηλαδή η ολοκλήρωση εσωτερικής αγοράς και η υποστήριξη περιφερειακής πολιτικής, οι δύο αυτές συνιστώσεις δεν ε, την χάνουν ολοκλήρωσης ή αλληλοσυσχετισμού. Και εμείς τονίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, διότι υπάρχουν μεγάλα χάσματα ως προς την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ενδοκινοτικά. Και αυτό αφορά για τα, κράτη, τα μελη που έχουν προσχωρήσει πιο πρόσφατα. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν συγκρίνουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέρον στο τομέα εκπαίδευσης, υγείας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ζητημάτων, μεταξύ βόρειων χωρών και ορισμένων νοτίων χωρών, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι δραματική και κυριολεκτό. Αυτές οι διαφορές μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει πραγματικά ολοκλήρωση των οικονομιών μας. Ένα σαφές παράδειγμα είναι οι τηλεπικοινωνίες. Ένα από τα μικρά προγράμματα τα οποία αναλύσαμε αφορά την χρηματοδότηση των, της ευρυζωνικότητας της ευρυζωνικής ψηφιακής επικοινωνίας σε ορεινές περιοχές. Ας πούμε στην Ελλάδα, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε εδαφική συνεργασία χωρίς να μετακινούνται οι άνθρωποι, τότε θα πρέπει να μετακινηθεί η πληροφόρηση. Αλλά για να κινηθεί η πληροφορία με υψηλή ταχύτητα χρειάζεται ευρυζωνική επικοινωνία, ακόμα και εκεί όπου οι αγορές δεν παρέχουν αυτή, αυτές τις υποδομές. Γιατί δεν υπάρχει ε, ε, βραχυχρόνιο κέρδος. Αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά πέρα από τις τηλεπικοινωνίες, οι διαφορές εδώ δεν αφορούν μόνο τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο 15 ή τις χώρες που προσχώρησαν μεταγενέστερα. Αφορά και το επίπεδο των 15. Ο περιβαλλοντικός τομέας είναι ένας άλλος τομέας όπου οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος παρουσιάζουν μεγάλα κενά σε σχέση με, τα, σε σχέση με τις αστικές περιοχές και μη. Η βιώσιμη ενέργεια είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτό αναφέρθηκε και από τον Επίτροπο σήμερα το πρωί. Μιλάμε για τους στόχους του 2020 και ένα μέρος αυτών των στόχων σε, σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αδύναμος συσχετισμός μεταξύ προγραμματισμού σε περιφερειακό επίπεδο και ευρωπαϊκής προοπτικής για την επίτευξη των στόχων του 2020 και δεν θα με εξέπλητε καθόλου εάν κατά τα επόμενα δέκα έτη δεν θα είμαστε σε θέση να ε, οδηγήσουμε στη σύμπλευση αυτών των δύο συνιστοσών όπως έγινε και με την έρευνα και την ανάπτυξη. Και δεν θα φτάσουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε μόνο ρυθμιστικές πολιτικές από τη μία πλευρά όπως γίνεται στην αγορά ενέργειας και από την άλλη πλευρά τα διαρθρωτικά ταμεία χωρίς σαφή συντονισμό, αυτό δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του 2020. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη ε, δυστυχώς τα χρώματα δεν φαίνονται καθαρά, δεν είναι και τα σωστά εδώ στη διαφάνεια. Τα σωστά χρώματα θα τα βρείτε στην έκθεση καθεαυτή. Θα ήθελα η Σίλβια να, βρει, να μου βρει τη σελίδα ή μπορείτε, ε, έχετε μία εκτύπωση των διαφανειών όπου εκεί τα χρώματα φαίνονται είναι τα σωστά. Αυτό είναι ένας τρόπος για να έχετε μία συνοπτική εικόνα των διαφορών στη, ως προς την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τις κοινωνικές υποδομές. Βλέπετε τις πράσινες περιοχές, τις κίτρινες και τις κόκκινες ή πορτοκαλί όπου το κόκκινο και το πορτοκαλί αποτελούν ανησυχητική κατάσταση και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μπορείτε να βρείτε τα σωστά χρώματα στην εκτύπωση των διαφανειών. Εδώ μιλάμε για τον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, η επόμενη διαφάνεια, και θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. Τώρα τι γίνεται σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και πώς υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εδώ βλέπετε ότι ότι έχουμε αποπειραθεί να δώσουμε πληροφορίες για τα διαρθρωτικά ταμεία και για τις ανάγκες υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε περιφερειακό επίπεδο, εθνικό και περιφερειακό. Και εδώ έχετε τις ποσοστίες αναλογίες της κατανομής του ΕΤΠΑ αναχώρα στις, ε, στον πρώην και νυν προγραμματισμό σε αυτές τις περιόδους ε, προγραμματισμού και βλέπετε ότι ένα 60 με 70% των διαρθρωτικών ταμείων ε, χορηγούνται για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στα νέα κράτη, ενώ η ποσοστία αναλογία είναι πολύ χαμηλότερη σε, στις χώρες ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Υπάρχουν όμως ορισμένες διαφορές. Βλέπετε για παράδειγμα ότι η Γαλλία δαπανά το τμήμα των διαρθρωτικών που τους απονέμεται περισσότερο για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος παρά, ε, παρά ό,τι κάνει, σε αντίθεση μάλλον με αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε, στα επόμενα στοιχεία. Στις επόμενες διαφάνειες έχετε ε, μία ε, κατανομή ανατομέα αυτών των πληροφοριών και βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες, δηλαδή ορισμένες χώρες αποφάσισαν ε, βάσει διαρθρωτικών να ε, ορίσουν ορισμένες προτεραιότητες. αποφάσισαν να φτάσουν σε αυτά αποτελέσματα χωρίς να γίνει διάχυση των διαρθρωτικών ταμείων σε πολλές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και επέμειναν σε ορισμένους τομείς. Εδώ έχετε τηλεπικοινωνίες, κοινωνικές ε, υποδομές, περιβάλλον και ενέργεια. Ε, γίνεται λόγος για εκατομμύρια ευρώ. Ίσως όμως θα ήταν σκόπιμο να δούμε το κατακεφαλήν εισόδημα για να δούμε ποιες είναι και οι προτεραιότητες των κρατών μελών. Δηλαδή ευρώ ανακεφαλή, να το δούμε έτσι διότι έτσι γίνεται και η απορρόφηση των ε, κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Και εδώ βλέπετε το μέρος των κονδυλίων που αφορά την διασυνοριακή συνεργασία για αυτές τις πέντε ευρείες κατηγορίες διαρθρωτικών. Και όπως βλέπετε, στην ε, τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού υπάρχει αύξηση, σαφής αύξηση στην χρήση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων για την διασυνοριακή συνεργασία. Άρα φαίνεται σαφές από τα στοιχεία αυτά ότι οι ανάγκες υπάρχουν, τα διαρθρωτικά ταμεία καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Το ζήτημα όμως είναι κατά πόσο υπάρχει επιτυχία στην χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για να πληρωθούν τα κενά. Υπάρχουν καλά νέα και τα βλέπετε σε αυτή τη γραφική παράσταση. Σε αυτή τη γραφική παράσταση, στην, ε, στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία σε σχέση με τη χρήση α, ανακατοίκους και εγκάρσια βλέπετε τις υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος όπως χρησιμοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ μας ε, λέει η γραφική παράσταση, μας δείχνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία με, εθνικές, ε, με βάση εθνικές μεταβλητές και παραλλαγές ε, μεταβαίνουν, γίνεται χρήση τους εκεί όπου υπάρχουν πραγματικά ανάγκες. Δεν θα πρέπει να σας εκπλήσουν τα αποτελέσματα. Είναι όμως ε, καθησυχαστικά, γιατί η σημασία αυτής της γραφικής παράστασης ε, δείχνει ότι ο μεγαλύτερος όγκος των διαρθρωτικών κονδυλίων υποστηρίζουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεμονωμένα προγράμματα είναι καλά, κατά ανάγκη, ή ότι κάποια χώρα δαπανά καλά τα χρήματα, οπωσδήποτε, αλλά σημαίνει ότι υπό ευρωπαϊκή ε, προοπτική ο αρνητικός συσχετισμός μεταξύ πρικοδότησης και κατανομής ε, ε, αποτελεί ένα σημαντικό και καλό νέο. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από αυτή την μελέτη υποστηρίζουν την ιδέα άμεσου συσχετισμού μεταξύ παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και της ε, πλήρωσης του στόχου, του κοινωνικού στόχου. Και αυτός ο συσχετισμός είναι ακόμα πολύ πιο ε, μεγάλος από αυτόν που θεωρούν τα θεσμικά όργανα ή κυβερνήσεις. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στα συμπεράσματά μας και τις συστάσεις. Έχουμε επτά σημεία που θα θέλαμε να σκεφτείτε. Καταρχήν, ότι η Ευρώπη αποτελεί μια περιφέρεια του κόσμου με μεγάλες διαφορές ως προς το επίπεδο και ποιότητα παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Αυτό οι διαφορές αφορούν κυρίως το χώρο. Και οι διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των ΙΠΑ. Αν δείτε την ε, ε πέμπτη έκθεση συνοχής, έχετε ορισμένες ενδιαφέρουσες χαρτογραφήσεις όπου η ευρωπαϊκή διάσταση συγκρίνεται με την αντίστοιχη των ΙΠΑ ως προς τη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Στις ΙΠΑ, η ΗΠΑ είναι μια περιφέρεια του κόσμου με, με, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των πολιτών εξαιτίας ε, διαφορών εισοδημάτων, φιλετικών διαφορών και ευκαιριών. Και πολλές φορές Ανησυχούμε ιδιαίτερα και η παρούσα κυβέρνηση των ΙΠΑ ανησυχεί ιδιαίτερα ως προς αυτές τις διαφορές μέσα στη ΣΥΠΑ. Αλλά ως προς διαφορές μεταξύ πολιτιών, οι ΙΠΑ παρουσιάζουν πολύ πιο ομοιογενή εικόνα σε σχέση με την Ευρώπη. Και αυτό σχετίζεται με την αξιοπιστία παροχής ε, υπηρεσιών και των ε, υπερεθνικών θεσμικών οργάνων. Εάν κανείς ε, καταφέρει αυτές τις πολιτικές με τόσο μεγάλες περιφερειακές διαφοροποίησεις, τότε υπάρχουν, υφίσταται ένα ουσιαστικό πρόβλημα, υπάρχουν εντάσεις. Άρα η επένδυση στις υποδομές υπό την ευρεία έννοια αποτελεί πρόκριμα για να ε, πληρωθούν αυτά τα κενά. Η δεύτερη υπόδειξη, η δεύτερη σύσταση είναι ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να είναι ε, σημαντική πτυχή αυτού του προγράμματος και δεν ενθαρρύνεται επαρκώς αυτή τη στιγμή από το παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Η πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο δεν βλέπουν να υπάρχει επαρκές αντιστάθμισα, αντιστάθμισμα, με συγχωρείτε, έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία με περιφέρειες άλλης χώρας. Αυτό σημαίνει όμως, σε μερικές περιπτώσεις, ότι χάνονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό σχετίστηκε με άλλες χώρες. Χτες ε, βρέθηκα σε μία συνάντηση στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο σε σχέση με ένα πρόγραμμα για την εξαγωγική διαδικασία και αξιολόγηση projects και ένας υπάλληλος μίλησε για επενδύσεις για τον καθαρισμό υδάτων ενός ποταμού που βρίσκεται κοντά στα σερβικά σύνορα για να ε, συμμορφωθούμε με την περιβαλλοντική νομοθεσία λοιπόν. Επενδύθηκαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ για τον καθαρισμό των υδάτων αυτού του ποταμού. Ο ποταμός Ρέι. 20 χιλιόμετρα, για 20 χιλιόμετρα και μετά Ισραήλ στη Σερβία, όπου υπάρχει μόλυνση υδάτων. Άρα ο αντίκτυπος στο περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή εκτός από ένα ε, μικρό μήκος 20 χιλιόμετρων, ε, όλα τα υπόλοιπα, σε όλα τα υπόλοιπα δεν γίνεται τίποτα. Τα 20 χιλιόμετρα δεν σημαίνουν τίποτα. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό χώρο, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για συμμόρφωση με τους κανονισμούς, θα πρέπει να μας απασχολήσει ο απότερος στόχος, τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μαζί με τις γείτονες χώρες, που είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια μέρα μπορεί να είναι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση. Το τρίτο συμπέρασμα ή σύσταση είναι ότι οι υποδομές είναι η απαρχή της ιστορίας, όχι το τέλος. Εάν υπάρχει ένα ε, χάσμα το οποίο δεν αντιμετωπίσουμε, εάν δεν υπάρχει έλεγχος, πραγματικός έλεγχος κυκλοφορίας ή εάν έχετε ένα νέο νοσοκομείο, ένα νέο σχολείο, αλλά τα διαρθρωτικά ταμεία απλώς χρηματοδοτούν και εποπτεύουν ως προς το, μια γέφυρα που χτίζεται ή ένα σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες. Πολλές φορές μπορούν οι ανάδοχες εταιρείες να αναλάβουν κάτι τέτοιο, αλλά με την κατάλληλη εποπτεία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά πώς θα ε, κλείσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ ε, ρυθμίσεων και κανονισμών που αφορούν την δαπάνη κονδυλίων, υποδομών και άλλοι, άλλες διαστάσεις ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν την παροχή καλών υπηρεσιών και προστασία των καταναλωτών. Τέταρτον, τέταρτη σύσταση. Κατά πόσο υπάρχει η κοινωνική δυνατότητα ανάληψης διότι πολλές φορές οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ε, απαιτούν από τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα τέλη έτσι ώστε να, καλυφθούν, να καλυφθεί το κόστος. Ή μιλάνε για συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να ε, λάβουμε τα κονδύλια. Όταν όμως ε, επαναδιαρθρωθούν τα δασμολόγια Πολλές φορές πολλοί δεν μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο. Αυτό βλέπουμε. Υπάρχει δηλαδή μία κοινή αυταπάτη. Δηλαδή παρέχουμε ένα νέο ηλεκτρικό δίκτυο, μιλάμε για την αύξηση των εισφορών ή των τελών και λέμε ότι ένα 15, οτι ότι 15-20% των τιμολογίων δεν θα πληρωθούν διότι τα τέλη δεν μπορούν να τύχουν κοινωνικής στήριξης. Και αυτό γίνεται διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η περιφερειακή πτυχή του θέματος σε σχέση με άλλες πτυχές. Πέμπτη σύσταση. Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Πρόκειται για την πέμπτη. Πρόκειται για το διακυβερνητικό επίπεδο διακυβέρνησης και ένα από τα ευρήματά μας είναι ότι αν δεν υπάρχει ε, εύρωστη πολιτική ηγεσία σε τοπικό επίπεδο, τότε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους δικαιούχους. Άρα τίθεται ένα θέμα διακυβέρνησης που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν αφορά τις Βρυξέλλες καθαρά. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το κατά πόσον οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να υποβοηθηθούν μέσα στα πλαίσια των δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξουν σε διοικητικό επίπεδο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με αυτές τις, σε αυτές τις προκλήσεις. Τέταρτη, έκτη με συγχωρείτε λέει μιλητής ε, σύσταση, τα ε, διαρθρωτικά ταμεία ως γενικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αυτό το θέμα ε, δεν είναι καθαρανομικό ή θεσμικό. Αφορά τμήμα του κοινωνικού μοντέλου, αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού μοντέλου. Διότι μιλάμε για προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας πρόσβαση στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Πρόκειται όμως για την ίδια γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί πρόκριμα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ε, διαφορές και τις ανισομέρειες. Τέλος, όλα αυτά δεν είναι εφικτά χωρίς μία σωστή προσαρμογή στην ιδιαιτερότητα των περιφερειών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσον αφορά το ευρυζωνικό στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας ή η, η επικοινωνία παθολόγων μεταξύ Λιθουανίας και Δανίας. Είναι κάτι που χρειάζεται τοπική υποστήριξη. Δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς της ε, χρηματοδότησης σε πραγματικά πολύ καλές υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτά τα project. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ εσάς όποιος επιθυμεί να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή και αξιόλογη. Βλέπει ορισμένες ε, καθαρές ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών και μέσα σε χώρες μέλη αλλά και διαφορές μεταξύ χωρών μελών κάτι που δεν μας εκφνιδιάζει βέβαια άλλωστε είμαστε σε εποχή λιτότητος και τα πράγματα μάλλον θα πάνε χειρότερα και όχι καλύτερα διότι πολλές χώρες μέλη μειώνουν τις ε, δημόσιες δαπάνες. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων των περικοπών και τα πράγματα θα χειροτερεύσουν σημαντικά. Δεύτερο, και συμφωνώ και εδώ με την παρουσίαση, η σημασία δηλαδή των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο και οι υπηρεσίες προσφέρονται στο ίδιο επίπεδο. Η ικανότητά τους λοιπόν να καινοτομήσουν, έστω και εν ώψη περικοπών των δημοσίων δαπανών, έχουν τη δυνατότητα ορισμένες περιφερειακές και τοπικές αρχές να βρουν νέες ιδέες για να εξασφαλίσουν ότι και στο μέλλον, μάλλον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον τα διαρθρωτικά ταμεία θα εξυπηρετούν ιδιαίτερα τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τέλος, υποδομή. Ορισμένες από τις συστάσεις αναφέρθηκαν στη σημασία της υποδομής. Συμφωνώ. Η συνθήκη της Λισαβόνας, ή μάλλον η ατζέντα της Λισαβόνας, δείχνει εν τέλει ότι πολύ λίγα από τα χρήματα δαπανώνται στα διαφορετικά ταμεία. Τα περισσότερα πηγαίνουν για την ατζέντα της Λισαβόνας. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Έχετε εξετάσει την ισορροπία μεταξύ διαφορετικών ταμείων που δίνονται στην υποδομή και των κοντιλίων που δίνονται, για παράδειγμα, στην οικονομία της γνώσης και ποια ισορροπία θα πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ, Σοφή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε για την ποιοτική εργασία και την ποιότητα της εκθέσεώς σας, την οποία θα μελετήσω προσεκτικά, διότι με έχει, μου έχει αναθέσει η Οικονομική Επιτροπή ε, τη σύνταξη μιας νομοδότησης για την καθολική υπηρεσία, καθώς επίσης και για την οδηγία ε, των υπηρεσιών οι υπηρεσίες καθολικού ε, ενδιαφέροντος λοιπόν είναι σημαντικές γιατί συζητούνται σε πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το πρόβλημα της ε, Γενικής Καθολικής Υπηρεσίας, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, είναι ότι ο ορισμός της υπηρεσίας αυτής είναι δύσκολος, αφού άπτεται και πολλών εθνικών ευαισθησιών. Δεν έχουμε όλες, ε, ούτε τους ίδιους οργανισμούς ε, δημοσίου συμφέροντος στις χώρες μας, ούτε και την ίδια νοοτροπία. ούτε άλλωστε συμμεριζόμαστε τις ίδιες σκέψεις ό,τι αφορά την κοινοπραξία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα το θέμα. Για παράδειγμα, στην χώρα μου, τη Γαλλία, το θέμα διαχειρίσεως των νερών ανατίθεται συστηματικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Άρα, επιτελείται δημόσια υπηρεσία από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ αλλού ε, είναι κάτι τέτοιο αδιανόητο. Υπάρχει λοιπόν μια περιπλοκότητα ε, των θεμάτων που πρέπει να αναλυθεί ώστε να περάσουμε μετά σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και πάντως πρέπει να αναλυθεί πριν να σκεφτούμε μια, πριν να αναλογιστούμε μια οποιαδήποτε τέτοια κοινή ευρωπαϊκή στάση. Ευχαριστώ. Μάτουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και για την ποιότητα των δεδομένων που μας υποβάλατε σήμερα. Αυτό αποτελεί μια πραγματική πρόκληση και αυτές οι υπηρεσίες θα μας απασχολήσουν κατά πολύ από τούδε και στο εξής. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά θα πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη διασυνοριακή συνεργασία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είχα την ευκαιρία να ε, εργαστώ άμεσα όταν η Ρουμανία δεν ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μετά την ε, προσχώρηση είχαμε συνεργαστεί με την ε, Ουγγαρία και τη Σερβία τότε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και αυτή τη στιγμή να γίνει αυτός ο συντονισμός που μας ε, υποδείξατε πολύ καλά. Σε σχέση με αυτές οι υπηρεσίες, θα ήθελα να πω ότι όταν έρχομαι ε, εδώ από τη Ρουμανία θα πρέπει να διανύσω έξι χώρες. Δεν υπάρχουν πια σύνορα και ούτε καν συνειδητοποιούμε ότι περνάμε τα σύνορα όταν τα περνάμε. Όμως αυτό που σας δείχνω μας δείχνει ότι έχουμε περάσει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Δείχνει ο μιλητής στο κινητό του. Πώς ε, θεωρείτε ότι μπορεί να ισχύσει ένα ενιαίο τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και εγώ μένω λίγα χιλιόμετρα ε, μετά τα σύνορα και πολλές φορές η περιαγωγή είναι πολύ κακής ε, ποιότητας και πολλές φορές ε, χρησιμοποιούμε παρόχους άλλων κρατών όπου τα τέλη που καταβάλουμε είναι 8 με 10 φορές υψηλότερα από ό,τι στη χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να επιληθεί και αυτό το θέμα της περιαγωγής και να ισχύει ενιαίο τέλος. Very much. Ε, ευχαριστούμε πολύ, Κατρίν. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε που ήρθαμε καθυστέρηση, αλλά ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Ίσως να το θίξατε το θέμα αυτό στην αρχή της ομιλίας σας, κύριε. Αλλά ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζω ως Ευρωβουλευτής όταν επισκέπτομαι την εκλογική μου περιφέρεια και με ρωτούν για χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου λένε κάθε φορά και μιλώ τώρα για τοπικές αρχές αλλά και άλλους κάθε φορά που έκαναν προσπάθεια να επιτύχουν κοινοτική χρηματοδότηση τραβάνε τα μαλλιά τους κυριολεκτικά και λένε ότι απελπίστηκαν και σταματούν και μιλώ τώρα και για το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν τις ικανότητες ούτε να εντοπίσουν ακριβώς τις ανάγκες τους, ούτε να τις ποσοτικοποιήσουν, να τις αναλύσουν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, καταλαβαίνω αυτό που έχετε ε, γράψει εδώ, είναι πού πάνε τα λεφτά. Αλλά εξετάστηκε για ποιο λόγο δεν υποβάλλονται τις χρηματοδότηση εν τέλει. Ε, Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Ήταν απόλυτα σαφής και αυτά που αναφέρατε είναι τροφή για σκέψη. Ως προς τις τηλεπικοινωνίες, θα ήθελα να σταθώ σε αυτή την ε, πτυχή. Είπατε ότι σήμερα θα πρέπει να κινείται η πληροφορία πολύ πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Η χαρτογράφηση, ο χάρτης μας ε, ε, που υπάρχει σελίδα 78 μας δημιουργεί ανησυχίες γιατί στο τομέα των ε, τηλεπικοινωνιών, στις μεταφορές και στην ε, κοινωνική, στις κοινωνικές υποδομές, τα στοιχεία είναι παρόμοια. Ιδιαίτερα για την ευρυζωνικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 αφορά τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, περνάει μέσω των άλλων χωρών στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ευρυζωνικότητα ως τομέα που θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ως προτεραιότητα. Παρά να υπάρχει διάχυση και να μην μας απασχολεί αυτός ο τομέας, διότι αυτός θα είχε μεγάλη επίπτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και αφορά και τη στρατηγική του 2020. Μιλάμε για νέες δεξιότητες, για νέα επαγγέλματα. Αυτό αφορά και την κοινωνική επικοινωνία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, βελτιώνοντας τις τηλεπικοινωνίες, πολλά μπορούν να επιτευχθούν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αν δούμε αυτές τις γραφικές παραστάσεις, αυτά τα διαγράμματα, βλέπουμε ότι το επίπεδο τηλεπικοινωνίας είναι πολύ χαμηλό. Είπατε ότι στις ΗΠΑ υπάρχει καλύτερος, ε, καλύτερες υποδομές και αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό περισσότερο. Και εγώ θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. Και ένα σχόλιο επίσης. Μιλείτε για τα διαφθορτικά ταμεία. Αυτό όμως που πραγματικά εννοείται είναι η πολιτική συνοχής και η αξία των διαφθορτικών ταμείων στο πλαίσιο αυτό δεν είναι μοναχά η χρηματοδότηση που προσφέρουν, αλλά και ο μηχανισμός προσφέρει η πολιτική συνοχής ώστε να διεξαχθεί αυτή η πολιτική να προσφέρει δηλαδή τις ε, δημόσιες υπηρεσίες έχοντας και ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό φροντίζοντας έτσι για την προσέγγιση στους πολίτες, στους εταίρους που συμμετέχουν στην πολιτική αυτή, στην εφαρμογή της, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και έργων και βέβαια ενισχύοντας και αυτό το διαμεθοριακό, διαμεθοριακό χαρακτήρα των πολιτικών. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Το σχόλιο μου έχει ως στόχο να δείξει ότι δεν είναι μοναχά η χρηματοδότηση εν προκειμένου, αλλά είναι πραγματική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία με την παροχή αυτή δηλαδή ε, υπηρεσιών καθολικού ε, ενδιαφέροντος και που είναι και από τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η ερώτηση που θα σας κάνω είναι η εξής. Ενδιαφερόμαστε πολύ για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής και των χρηματοδοτικών μηχανισμών της. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εμπόδια στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της ε, πολιτικής προέρχονται από άλλους τομείς της ευρωπαϊκής δραστηριότητας και τα κολλήματα αυτά, οι φραγμοί αυτοί που εξακολουθούν να υπάρχουν και μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς καθιστούν την πλήρη χρήση, την πλήρη εκμετάλλευση της πολιτικής συνοχής για την παροχή δηλαδή υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος πιο δύσκολη. Ερώτηση. Εξετάσατε και αυτούς τους φραγμούς που, από τους οποίους είναι γεμάτη η ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά την ε, προσφορά από την πολιτική συνοχή υπηρεσιών καθολικής, καθολικού συμφέροντος. Για παράδειγμα, νοσοκομεία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πραγματικά σε παραγωγικές περιοχές. Η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν μπορεί να περάσει από την άλλη των συνάωρων λόγω αυτών των φραγμών που η ενιαία αγορά ακόμα δεν έχει ε, καταργήσει. Βρίσκεται λοιπόν τέτοιου φραγμούς και άλλους που καθιστούν δύσκολη την προσφορά ε, υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος. Τα έχετε εξετάσει αυτά. Δεύτερη ερώτηση τώρα σε ό,τι αφορά την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος για τις οποίες μιλούμε. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει περάσει και στον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές σε ό,τι αφορά και την ποιότητά τους και την προσβασιμότητά τους από πλευράς του κοινού. Έχετε εξετάσει και τον ρόλο αυτό της τεχνολογικής αλλαγής, της αλλαγής των μηχανισμών της προσφοράς καθολικής υπηρεσίας, γιατί για το μέλλον η πολιτική συνοχής μπορεί να προωθήσει και την αλλαγή της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την ερεσιμότητα την επιβολή όρων δηλαδή για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τέτοιες υπηρεσίες. Διερωτώ με αν τα έχετε εξετάσει αυτά Συνεχισή σας. Δεν βλέπω τώρα άλλες ή άλλους συναδέλφους να επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ευχαρίστως λοιπόν αν θέλετε να απαντήσετε εσείς ή οι συναδελφοί σας. αναθέτουν σε μένα οι συναδελφοί μου την ευθύνη να κάνω οποιοδήποτε λάθος ενδέχεται να κάνω. Τα σχόλια λοιπόν, αναπόφευκτα θα είναι κάπως πιο προσωπικά, διότι ορισμένες από τις ερωτήσεις ε, υπερβαίνουν και τα όρια της ίδιας της μελέτης. Θα αρχίσω με το σημαντικό ερώτημα σχετικά με τις εθνικές παραδόσεις, τις οποίες εγώ θα διασυνδέσω και με το τελευταίο σχόλιο της κυρίας Χίπνερ. Λοιπόν, ναι, όλοι έχουμε διαφορετικές παραδόσεις και νομικούς φραγμούς για την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Όμως, ας επανέλθουμε στο παράδειγμα της e-Baltic Cooperation, της ηλεκτρονικής συνεργασίας βαλτικών χωρών με ορισμένες σκανδιναβικές όπως Δανία, Σουηδία και βέβαια από την άλλη μεριά μερικές από τις ε, πρόσφατα ενταχθήσεις βαλτικές χώρες όπως Λετωνία ή Λιθουανία. Το θαύμα είναι ότι επέλυσαν τα προβλήματα αυτά. Σας εξηγώ το πρόβλημα. Εάν έχετε ρυθμίσεις που απαγορεύουν έναν γιατρό στη Λιθουανία να κάνει μια διάγνωση για λογαριασμό ενός ασθενούς στην Δανία δεν θα μπορούν να γίνονται και ανταλλαγές ηλεκτρονικών αρχείων των ακτινολόγων για να συμβάλλουν στην ε, διάγνωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι προσπάθησαν και το έλυσαν το πρόβλημα αυτό. Πώς το έκαναν, όχι με σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία, αλλά με συγκεκριμένες ειδικέ συμφωνίες μεταξύ των αρχών υγείας με τον των χωρών μελών. Και λειτουργήσε ο τρόπος αυτός. Να λοιπόν μια ενδεχόμενη επιλογή εκ των κάτω. Μια προσέγγιση λοιπόν από τα κάτω όπου η πολιτική συνοχής προσφέρει οικονομικά κίνητρα για να γίνουν αυτά τα πράγματα και να ε, δώσει όθηση στους ανθρώπους να κάνουν τους απαραίτητους συνδυασμούς των προσπαθειών τους. Χρήση λοιπόν της πολιτικής συνοχής και των διαφορετικών ταμείων ως εργαστήρι για τον συνδυασμό αυτών των διαφορετικών εθνικών παραδόσεων και μέσα σε μια αναπτυξιακή προοπτική στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο όπου ίσως μετά από δεκαετίες βέβαια, θα μπορούμε να αντισταθούμε στα, στις δοκιμασίες στρες και να υπάρχει μια επιτυχία σε μια πιο ανοιχτή κοινωνία. Βέβαια, δεν νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν με μια προσέγγιση εκ των κάτω. Από τη σκοπιά αυτή Εξακολουθεί νομίζω να υπάρχει ένα είδος ελίποντος κρίκου μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών ε, πολιτικών όπως της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών άλλων τομέων σε άλλους τομείς. Το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα της περιαγωγής. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό είναι καλό, διότι όπως θα γνωρίζει η Κομισιόν, κάποια στιγμή έλαβε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την περιαγωγή, το roaming, διότι ανακαλύψαμε εν τέλει ότι μετά από πλήρωνες οδηγίες που ζητούσαν το άνοιγμα της αγοράς για την κινητή τηλεφωνία, έγινε ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν και πριν από την απόφαση της Κομισιόν. Ο, το ιδιωτικό τέλος που λάμβαναν οι εταιρείε της τηλεφωνίας κάθε φορά που εσείς διαβαίνατε τα σύνορα δεν είχαν όρια. Κάποια στιγμή λοιπόν η Κομισιόν έλαβε καθαρά μια απόφαση εκ των άνω να βάλει μια οροφή σε αυτά. Όχι να καταργήσει τις διαφορές, αλλά να τους βάλει μια οροφή και να προστατεύσει έτσι τους καταναλωτές. Πώς τώρα συνδυάζεται αυτό με τη συζήτησή μας περί πολιτικής συνοχής. Το βλέπω ως απόδειξη του γεγονότος ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, και ο καλύτερος, ο ιδανικός ίσως είναι η Ευρωβουλή, όπου να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα ή κοινά οράματα για τα σημαντικά αυτά θέματα και να γίνει προσπάθεια συνδυασμού της πολιτικής συνοχής με τις άλλες πολιτικές της ε, ε, Κομισιόν. Όπως είπα στην αρχή της παρουσιάσεώς μου, ορισμένες φορές ευνηδιάζομαι, βλέποντας για παράδειγμα, πως η Γενική Διεύθυνση Ενίας Αγοράς διεξάγει περιορισμένο διάλογο με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Έστω και αν η πολιτική συνοχή σε ορισμένες περιπτώσεις στηρίζει τις κερφαλιοχικές επενδύσεις των επιχειρήσεων εκείνων που ελέγχονται από την Γενική Διεύθυνση Ενίας Αγοράς. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα αν από την αρχή οι διάφοροι κλάδοι των ευρωπαϊκών πολιτικών κάθονταν και συνομιλούσαν και έβαζαν όρους για την ίσπραξη κονδυλίων αυτή τη στιγμή πρώτα επιτευχθούν κάποια αποτελέσματα υπέρ των καταναλωτών. Καλύτερα έτσι, πριν να δώσετε τα λεφτά. Και όχι πρώτα να δώσετε τα λεφτά και μετά τα λεφτά και να δείτε μετά ότι στην ουσία χρησιμοποιούνται αυτά για να προστατεύσουν τις μάρκες της ε, επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι μονομικό θέμα, διότι από την άποψη τη νομική οι διαδικασίες ε, δημοσίων προμηθειών κτλ. θα πρέπει να γίνονται σεβαστές, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά στην ουσία είναι και ζήτημα ουσίας. Πραγματικού, ουσιαστικού περιεχομένου δηλαδή. Για το θέμα τώρα, βέβαια δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα σχόλια, αλλά δηλώνω πόσο ευχαριστημένο είμαι από αυτή την ζωηρή συζήτηση που διεξήχθη, αλλά ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι η σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης, της δημοσιονομικής κρίσης καλύτερα, και τη προσφορά καθολικών υπηρεσιών στα πλαίσια της πολιτικής συνοχή που δεν καλύπτεται από την παρούσα μελέτη. Ωστόσο, <clears throat> θα συστήσω θερμά στην παρούσα Επιτροπή να αναλογιστεί σχετικά με τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης και των περιορισμών που επιβάλλει που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο όλο το πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Όχι μόνο λόγω περικοπής κονδυλίων των ταμείων. και που οδηγούν και στην έλλειψη συγχρηματοδότησης από τις χώρες μέλη ή και ανεξάρτητα που οφείλεται και σε αυτό αλλά και λόγω της επιλογής έργων που δεν ακολουθούν πλέον προτεραιότητες της πολιτικής αλλά μάλλον λιγότερο σημαντικές οικονομικές προτεραιότητες. Δηλαδή τα έργα που πιο εύκολα χρηματοδοτούνται, για παράδειγμα από τον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν αυτομάτως προτεραιότητα, ακόμα και αν υπάρχουν και άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, που επειδή είναι πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθούν από ιδιωτικά κονδύλια, στην ουσία αναβάλλονται ή καταργούνται από τις χώρες μέλη. Και αυτό λοιπόν είναι θέμα κατεύθυνση τη διαδικασία από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών και προσπάθειας αποφυγής αυτού του παιχνιδιού ανάμεσα στα δημοσιονομικά, στις στα δημοσιονομικά πακέτα, ώστε η πραγματική στόχη της πολιτικής συνοχής εν τέλει να υπονομεύεται ή να παρακάμπτεται και να χρησιμοποιείται για άλλους στόχους. Μου έγινε και ένα σχόλιο σχετικά με αυτόν τον εφιάλτη της ε, απόκτησης χρηματοδοτήσεως από πλευρά των τοπικών αρχών. Αυτό δεν το έχουμε εξετάσει στη μελέτη, αλλά έχω ένα σχόλιο το οποίο σχετίζεται με τα όσα είπα στην αρχή της παρουσιάσεώς μου. Είναι λοιπόν σαφές ότι αν το μέλλον της πολιτικής συνοχής θα εξακολουθήσει να βασίζεται σημαντικά σε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην είναι απλώς θέμα μεταφοράς κονδυλίων από τον κοινοτικό στον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά να είναι και ένα πραγματικό δημιουργικό πείραμα και να περνάει από την ευρωπαϊκή διάσταση στην τοπική διάσταση. Θα συνιστούσα λοιπόν να δοθεί συνδρομή στις τοπικές αρχές για να λαμβάνουν χρηματοδότηση για, τα όσα, για τις πραγματικές τους ανάγκες και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μπει στους κανόνες του παιχνιδιού και άρα στους κανονισμούς. Διότι είναι προφανές ότι οι αρχές των μεγάλων αστικών κέντρων, των εύπορων περιφερειών, που έχουν εν τέλει λιγότερη ανάγκη στήριξης, είναι ωστόσο και πιο ικανές οι αρχές αυτές να υπερβαίνουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα συστήσω λοιπόν να επινοηθούν νέοι τρόποι ώστε να μπορέσετε να συνδιαλεχθείτε με τον δήμαρχο του μικρού χωριού στην, ή τον κοινοτάρχη ε, στη Ρουμανία ή στον νότο της Ιταλίας και να βοηθήσετε αυτό το συγκεκριμένο δήμαρχο να μεταφέρει τις ιδέες του σε συγκεκριμένα έργα και να λάβει τη χρηματοδότηση για την εκτέλεσή τους. Και το τελευταίο μου σχόλιο αναφέρεται στην σχέση που ανέπτυξε η κυρία Χύπνερ που νομίζω ότι έχει και προσωπικό ε, ιστορικό για να θυμάται ότι η πολιτική συνοχή δεν είναι μοναχά θέμα διαφθορτικών ταμείων. Δεν είναι μονάχα χρηματοδοτήσεις, είναι πολιτική. Και το σχόλιο μου είναι ότι ειδικά σε αυτές, στο τομέα αυτών των καθολικών υπηρεσιών, εγώ προσωπικά ως Ευρωπαίος πολίτης θα ήθελα πολύ στο μέλλον να είναι, να λάβει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα πολιτικής και λιγότερο απλής κατανομής ε, πιστώσεων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε στους λίγους εμάς που είμαστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους εμπειρογνώμονες που συνεργάστηκαν μαζί σας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μας, ιδιαίτερα συζητώντας για το μέλλον και τις προτεραιότητες καθώς και την αρχή της αιρεσιμότητας, της πολιτικής συνοχής και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μελέτη στο μέλλον. Λίγη αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και υπάρχει άλλο ένα θέμα που είναι η επόμενη συνεδρία, 26 και 27 Ιανουαρίου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλοι τη συνεδρία. ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ η Πρόεδρος και τους Διερμηνείς. Ευχαριστώ και οι Διερμηνείς.